Ε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση που είναι καθ' αφιερωμένη στην ανταλλαγή απόψεων με δύο υπουργούς της Δανίας, εκπροσώπους της Δανικής Προεδρίας. Τον Όλε Ζών και πρώτα τον Χένρικ Ντάμ που ήταν και πρώην Ευρωβουλευτής. Και κύριο Σώνα αν δεν καλά, ήταν πρώην Ευρωβουλευτής. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Δανό Πρωθυπουργό στην ε, Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας α, ε, τελειώσουμε όμως με το τσάι πρώτα. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη συναντηθεί ατύπως με τον Δανό Πρωθυπουργό. Εγώ το συνάντησα και στην Κοπεχάγη και είχα μια πολύ χρήσιμη συνάντηση με τον Χένρικ Ντάμ. Οπότε αν υπομονούμε να σε ακούσουμε, έχει το λόγο και Καλώς ήρθες και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το νέο σου ρόλο, τη νέα σου ιδιότητα ως Υπουργό Μεταφορών του Βασιλείου της Δανίας και ως ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ. Το επόμενο εξάμεινο η Δανία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου, κάτι που περιμέναμε με αδημονία. Γι' αυτό και σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερος που θα σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, με μεγάλη χαρά θα συζητήσω μαζί σε αυτό το πρόγραμμα. Ως πρώην Ευρωβουλευτής γνωρίζω ότι είναι πολύ σημαντική η στενή και επικοδομητική συνεργασία της Προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζω επίσης ότι το έργο των διαφόρων επιτροπών έχει αποφασιστική σημασία για να υλοποιηθούν οι στόχοι και οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Επιμένω στο γεγονός ότι η Δανία αντιλαμβάνεται πλήρως τις ευθύνες που επομίζεται η εκάστοτε Προεδρία και έχει πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει. Πάντως, ε, έχουμε έρθει πολλές φορές με τους συνεργάτες μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχω τακτικές επαφές με πολλά μέλη της Επιτροπής σας. Επίσης, έχω τακτικές επαφές και με τον πρόεδρο της Επιτροπής σας, τον Μπρά Σίμψον. Και για θέματα μεταφορών, η ιδανική, η ιδανική Προεδρία θα ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με ορισμένα ντοσιέ που της είναι προσφυλή. Ο συνάδελφος είναι αρμόδιος για θέματα ναυσιπλοείας και αργότερα θα σας παρουσιάσετε τα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές. Κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας θα έχουμε στις 23 και 24 Μαρτίου το πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών και στις 7 και 8 Ιουνίου το δεύτερο. Το θέμα θα είναι η οικολογική ανάπτυξη, η πράσινη ανάπτυξη και η διέξοδος από την οικονομική κρίση. Γιατί μόνο ένας αποτελεσματικός κλάδος μεταφορών θα μπορέσει να συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης από τα βασικά σημεία του προγράμματος της Δανικής Προεδρίας θα είναι η αναθεώρηση του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου, η αναθεώρηση του πακέτου για τα αεροδρόμια και η δημιουργία ή η προώθηση του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης του Γαλιλαίου. Σε ό,τι φορά την αναθεώρηση του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου, ευελπιστούμε σε συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί γνωρίζουμε ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντική για να ενισχυθεί η θέση του, των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Είναι μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ε, να θεσπίσουμε κοινούς ενιαίους ομοιόμορφους κανόνες για να μπορούν να να κυκλοφορούν τα τρένα ε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια, είναι δύσκολε οι εργασίε για το σιδηροδρομικό πακέτο, αλλά πιστεύουμε ότι θα έχουν αίσιο πέρα. Η αναθεώρηση του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου θα είναι πολύ σημαντικό βήμα για την ε, πρόοδο στην Ευρώπη, γιατί θα εξασφαλίσει καλύτερη λειτουργία των σιδηροδρόμων, κάτι που θα είναι προς όφελος και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις μεταφορές εμπορευμάτων και προς όφελος των επιβατών είχα την ευκαιρία να συναντήσω την Τώρα Σαρακίνη, την εκπρόσωπό σας και είχαμε καταπληκτική συνεργασία στην προσπάθεια να διεκπαιρεώσουμε από κοινό αυτό το σχέσιο. ό,τι αφορά τώρα την αναθεώρηση των κατευθύνσεων ε, για το σιδηροδρομικό πακέτο και το ΕΡΤΕ, θα είναι σημαντική προτεραιότητα της Ισοδανικής Προεδρίας και θέλουμε να ολοκληρώσουμε και αυτή την αναθεώρηση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την αγραστή συνεργασία που ξεκίνησε στον τομέα αυτό η Δανική Προεδρία, γιατί ξέρουμε ότι αναμένονται σκληρές εργασίες στο Συμβούλιο. Γιατί η αναθεώρηση των προσανατολισμών ε, αυτών είναι σημαντικός, σημαντική ε, απέτηση για την ευρωπαϊκή πολιτική. Θα πρέπει στηρίζοντας την εσωτερική αγορά, να επενδύσουμε περισσότερο στις υποδομές και να εξασφαλίσουμε καλύτερη διασύνδεση των χωρών της ευρωπαϊκής αγοράς. Επίσης, θέλουμε να, να συσφίξουμε τους ε, δεσμούς μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και να διαμορφώσουμε πρόσφορο έδαφος για τις διασυνοριακές επενδύσεις. Οι υποδομές είναι εκ κάνει προϋπόθεση και για την ανάπτυξη. Και με την πρόταση αυτή δημιουργούμε ένα καλύτερο δυναμικό ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία. Στόχος μας είναι να προβούμε σε μια γενική αναθεώρηση αυτού του θέματος και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η πρόταση με τον προπολογισμό που έχουμε προβλέψει. Γιατί υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί και θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε κάποιες νέες υποδομές, αλλά οι πόροι που έχουμε για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών υποδομών είναι απαραίτητοι για να καταλήξουμε στην, στις κατευθυντήριες γραμμές για την αναθεώρηση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Υπάρχει και το σχέδιο Connecting Europe Facility. Και αυτό το πρόγραμμα είναι σημαντικό και περιμένουμε τις συζητήσεις στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να γίνουν παράλληλα με την ε, ε, μεταρρύθμιση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να υποβάλουμε και την έκθεση πρόοδου για το Connecting Europe Facility. Πάντως θέλουμε οι δύο αυτές τις προτάσεις, το Connecting Europe και η μεταρρύθμιση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, να εγκριθούν από κοινού. Σε ό,τι αφορά τώρα το πακέτο για τους αερολιμένες, είναι μια ακόμη προτεραιότητα της Δανικής Προεδρίας, γιατί οι αερομεταφορές είναι ο δημοφιλέστερος τρόπος ε, μεταφοράς και ο πιο διαδεδομένος και μια εύρυθμη λειτουργία των αερομεταφορών ε, εξασφαλίζει καλύτερη σύνδεση των ευρωπαϊκών πόλεων. Θα πρέπει όμως το τομέας των αερομεταφορών να σέβεται και να προστατεύει το περιβάλλον. Θα πρέπει να ενισχυθεί το δυναμικό του, και η αποτελεσματικότητα του τομέα των αερομεταφορών, βελτιώνοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα και το επίπεδο των υπηρεσιών. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις και για τη μείωση του θορύβου και στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία για τη μείωση του θορύβου. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δορυφορικής πλοήγησης, το Γαλιλαίο, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρμόδια για το θέμα αυτό είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας, ήτρε, και για τα TNT, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, θα γίνουν διαβουλεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Πάντως είπαμε και στην Ήτρε ότι το Γαλιλαίο είναι προτεραιότητα της ε, Δανικής Προεδρίας. Θέλουμε ένα ε, πάγιο πλαίσιο για το Γαλιλαίο και μας ενδιαφέρει και μια οριζόντια, μια γενική προσέγγιση για το θέμα αυτό. Ωραία, ως προς τις οδικές μεταφορές. Η πρόταση της οδηγίας για τις οδικές μεταφορές είναι επίσης σημαντική. Στόχος της είναι η καλύτερη διαχείριση των οδικών μεταφορών, μια καλύτερη κατανομή του φόρτου ε, και θα προσπαθήσουμε και στον τομέα αυτό να σημειώσουμε πρόοδο. Ταυτόχρονα η, Γενική, η Ιδανική Προεδρία θα δώσει έμφαση σε τρία ακόμη σημεία. Στην διατροπικότητα, ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή αποτελεσματικότητα και στη μείωση των εκπομπών των καυσαερίων. Επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε τη διατροπικότητα στις ε, διάφορες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο ζήτημα που μας απασχολεί είναι η ασφάλεια στα αεροδρόμια. Γιατί οι διατάξεις περί ασφαλείας είναι όλο και πιο περίπλοκες και προβληματίζουν και τους εργαζόμενους και τις ε, αεροπορικές εταιρείες αλλά και τους επιβάτες χωρίς ταυτόχρονα να επιφέρουν προστιθέμενη αξία. Θα συζητήσουμε και τους κανόνες για το χρόνο ανάπαυσης των εργαζομένων, για τους πιλότους και το πλήρωμα. Χρειάζεται επαρκής χρόνος ανάπαυσης ε, για να μπορούν και οι πιλότοι και το πλήρωμα να διεκπαιρεώνουν το έργο τους ε, ε, σε καλές ηθίκες. Στις 17 Απριλίου θα διοργανώσουμε στη Δανία μία διάσκεψη για τη διαχείριση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Το σύστημα RTNS. Η συνδιοργάνωση εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Δανία είναι η πρώτη χώρα του κόσμου που, θα εφαρμόσει αυτό το σύστημα σε όλο το σιδηροδρομικό του δίκτυο πριν το 2021 και σε αυτή τη διάσκεψη θα προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων για το σύστημα αυτό. Μια άλλη διάσκεψη θα γίνει στις 24-25 Μαΐου για τη χρηματοδότηση των μεγάλων σχεδίων υποδομών και εκεί προβλέπεται συνδιοργάνωση Δανικής Προεδρίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συζητήσουμε μεγαλεπίβολα σχέδια υποδομών. Στην Δανία είχαμε πολλές εμπειρίες με τις μεταφορές. Έχουμε για παράδειγμα τη γέφυρα που συνδέει την Κοπεχάγη με το Μάλμε της Σουηδίας και τη σύνδεση Δανίας-Γερμανίας. Έχουμε πολύ χρήσιμες εμπειρίες ε, διασύνδεση και θα τις παρουσιάσουμε σε αυτές τις διασκέψεις. Επίσης, 27 Ιουνίου θα έχουμε μια διάσκεψη για το δικό δίκτυο, για τις οδικές μεταφορές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί πάλι θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για θέματα ασφάλειας στις μεταφορές. Ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για, τις για την ασφάλεια στις μεταφορές. Σε ό,τι αφορά την σωστή παιδεία α, για, τις... για την κυκλοφορία και εκεί έχουμε εμπειρία στην Δανία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την άσκηση της Προεδρίας. Ε, έχουμε επίγνωση του δύσκολου έργου που μας περιμένει, αλλά πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα και των μεταφορών και των υποδομών, ώστε να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με του ε, ομιλητέ από τι ομάδε. Ο κύριο Γκρό είναι πρώτο. Δεν θα σα αναφέρω όλα τα ονόματα τώρα. Δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ. Καταρχάς, καλή επιτυχία. Και σε εσά και στου συνεργάτε σα. Έχετε πολλά στον τομέα των μεταφορών να κάνετε. Ελπίζω μετά από έξι μήνε να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σύντομα, Νομίζω στην αναδιατύπωση το Κοινοβούλιο ε, τόνισε πολύ συγκεκριμένα ένα σημείο, το ρόλο δηλαδή του ρυθμιστή στις διάφορες χώρες. Ε, αφήσαμε τα άλλα θέματα για να σας δώσουμε την ευκαιρία να κλείσετε το θέμα αυτό. Και τα κρατημέλη βεβαίως πρέπει να πιστούν ότι εμείς ε, θέλουμε να έχουμε ένα, μια ανοιχτή αγορά και καλώς ρυθμισμένη. Αν λοιπόν μπορούμε να μπορείτε να συμφωνήσετε με το Συμβούλιο ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε το σημείο αυτό, νομίζω ότι τα υπόλοιπα δεν θα καταρρεύσουν για λεπτομέρειε. Τώρα, για, τις, ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα θέλουμε να προχωρήσουμε, γιατί οι επενδύσει αυτή τη χρονική στιγμή ε, μπορεί να μην είναι στην ημερήσια διάταξη όλων των χωρών, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μέσο οι επενδύσει για να φύγουμε από την, ε, από την κρίση αυτή. Η πιλωτική φάση λοιπόν υπάρχει αρχικά, αλλά δεύτερον πρέπει να δούμε και ποια είναι τα, τα κίνητρα για, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Θα πρέπει αυτό να συνδεθεί με συγκεκριμένε αποφάσει. Ελπίζω ότι σε κάθε περίπτωση ε, και εσεί όπω και εμεί θα κάνετε τη δουλειά σα και η Κομισιόν δηλαδή θα βρει μια ισορροπία μεταξύ ε, ε, μεταφορών, περιφερειακή πολιτική που επίση έχει να παίξει μεγάλο ρόλο ε, στι στις μεταφορέ και δεν θα μιλούμε θεωρητικά για του επόμενου έξι μήνε χωρίς να ε, δίδονται συγκεκριμένες ε, αποφάσεις. Οπότε είμαι της ε, άποψης ότι από το Συμβούλιο θα πρέπει αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα της ετοιμότητας, της διαθεσιμότητας που δείχνουμε για να τα λύσουμε, θα πρέπει να τα τονίσετε έτσι ώστε να μην ξεκινήσουμε να κάνουμε ατέρμονες συζητήσεις θεωρητικές. Τώρα για το πακέτο για τα αεροδρόμια για μας ε, συζητήθηκε σήμερα το πρωί, τονίστηκε επαρκώς. Θεωρούμε ότι η αναγκαιότητα ενός τέτοιου μέτρου θα εξαρτηθεί από το, από το κατά πόσο θα ωφελήσει τους χρήστες. Ελπίζουμε να φέρει πιο πολύ ασφάλεια, ελπίζουμε να φέρει καλύτερη ε, ε, ποιότητα υπηρεσιών. Και ελπίζουμε αυτή η, η θεωρία και η θεωρητική συζήτηση που έχουμε κάνει να μεταφραστεί και σε έργα. Ξέρετε ότι το 2012 είναι ένα πολύ σημαντικό έτος Υπάρχουν και τα functional air blocks, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Ε, και βεβαίω πρέπει να δούμε τι γίνεται και σε κάθε κράτο μέλο. Τα κράτη-μέλη έκαναν ε, πολλά για να φτάσουν στο σημείο αυτό. Οπότε τώρα επαφιέται στα χέρια τη ε, Προεδρία του Συμβουλίου. Ελπίζουμε τα θέματα αυτά να προωθηθούν, έτσι ώστε το, το τέλο του 2012 να έχουμε κάνει ένα βήμα προ τα εμπρό. Οπότε ρωτώ, στην χώρα σα τι σκέφτεστε να κάνετε για το θέμα αυτό συνολικά. Πώ σκέφτεστε να συμβάλλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλκαντράουι από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου, τον Υπουργό για την εισαγωγή που μας έκανε. Έχετε μπροστά σας μια έντονη περίοδο εργασίας. Εξάλλου, οι τελευταίε προεδρίε άνοιξαν κάποιου φακέλου πολύ σημαντικού και σα ευχόμαστε καλή τύχη. Ε, μιλήσαμε για την ε, οικονομική πολιτική και η πολιτική μεταφορών μπορεί να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη. Είναι σημαντικό λοιπόν σε συνθήκες κρίσης να μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει το θέμα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και του ταμείου που προβλέπεται για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι η Δανέζικη Προεδρία θα τολμήσει και θα είναι θαραλέα και απέναντι στους συναδέλφους της στο Συμβούλιο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει σύγκρουση με το Συμβούλιο για μια σειρά από κρίσιμα σημεία ήδη. Μιλάω για την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό των διευρωπαϊκών δικτύων ε, μεταφορών, ε, για τους όρους, τις προϋποθέσεις που θέλουμε να επιβάλλουμε εμείς δεν θέλουμε δηλαδή να δώσουμε λεφτά στα κράτη-μέλη για να υλοποιήσουν τις υποδομές. Τις δίνουμε με κάποιες προποθέσει. Δηλαδή αν υπάρχουν ε, έργα με υπεραξία ευρωπαϊκή, προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν ε, ως προς την τεχνική διατροπικότητα και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός ε, αυτών των διαφορετικών μορφών μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίση δεν θα πρέπει αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιούνται για σκοπού μη Ευρωπαϊκού. Αν χρησιμοποιηθούν ποτέ έτσι θα πρέπει να επιστραφούν για να χρησιμοποιηθούν για του σκοπούς που θέλουμε εμεί, δηλαδή για έργα πάντα με ευρωπαϊκή διάσταση. Είναι σημαντικό να υπάρχουν επίση επαρκεί οικονομικοί πόροι, στην πρόταση τη Κομισιόν όμω για το Connecting Europe Facility, υπάρχουν 31,7 ε, δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται. Ελπίζω να καταφέρετε να πείσετε τους συναδέλφους σας ε, στο Συμβούλιο ε, να διατηρηθεί αυτό το ποσό που είναι οπωσδήποτε απαραίτητο για να υπάρξει πρόοδος. Σε εσά δηλαδή αφινόμαστε εμείς, θεωρούμε ότι θα έχουμε την υποστήριξή σας. Επίσης το πακέτο για τα αεροδρόμια και γενικά τις αναέριες μεταφορές. Είναι σημαντικό που η Κομισιόν, και σωστό που η Κομισιόν θέλει να μεταρρυθμίσει τον τομέα αυτό με διάφορε πρωτοβουλίε. Τις πρωτοβουλίε αυτέ θα τις ε, μελετήσουμε μεγάλη προσοχή και θέλουμε να προστατεύσουμε πάντα τον καταναλωτή παύλα ε, επιβάτη που συχνά βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Σε ό,τι αφορά τη δική μου ομάδα του σοσιαλιστές, εμείς είμαστε υπέρ ενός αυτόματου περάσματος του προσωπικού από τη μία επιχείρηση στην άλλη όταν αλλάζει ο πάροχος, όταν αλλάζει η εταιρεία. Δεν θα πρέπει να απολύονται οι παλιοί εργαζόμενοι. Και επίσης, όπως είπε ο Μάθιου Γκρός, είναι σημαντικό να τονίσουμε το εξή. Αν εμείς θέλουμε να έχουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών, θα πρέπει να μην ξεχνάμε και τον, ευρωπαϊκό, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και θα πρέπει να υλοποιήσουμε τις συμφωνίες τις οποίες έχουμε συνάψει και εσείς ως Προεδρία φυσικά έχετε την ευθύνη να συνοδεύσετε αυτή την προσπάθεια, για να το πω έτσι, αυτή τη δέσμευση που έχουμε να αναλάβει, ούτως ώστε να σημειωθούν σημαντικά βήματα μέσα στο 2012. Αυτά για μας είναι τα πιο σημαντικά θέματα επί των οποίων πρέπει να εργαστούμε. Ακόμα μια φορά καλή τύχη και βασιζόμαστε σε εσά για να επιλύσουμε οποιαδήποτε προβλήματα. Ο κύριος Ουτζίας από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Μας παρουσιάσατε ένα πρόγραμμα που είναι και πρακτικό, αλλά και φιλόδοξο παράλληλα. Πρακτικό γιατί θέτει στόχους υλοποιήσιμους και φιλόδοξο γιατί για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους αυτό σημαίνει για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι πρέπει να κάνουν έτσι μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είσαστε, ήσασταν ευρωβουλευτή στο παρελθόν και να σας πω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν προχωρούν αναεξάμεινο, μετά πηγαίνουν, φτάνουν στο μηδέν και ξαναρχίζουν από το μηδέν. Συνεχίζουν από εκεί που είχαν μείνει το προηγούμενο εξάμεινο. Θα ήθελα λοιπόν και στον τομέα των μεταφορών να βάλετε ε, τον ίδιο ενθουσιασμό ε, και για τους φακέλους ε, που δεν έχουν κλείσει ακόμα στις προηγούμενες προεδρίες. Δηλαδή, αν όμως εσείς δείξετε ζέση, τη ζέση την απαραίτητη, μπορείτε να τα προχωρήσετε αυτά τα θέματα. Ιδίως, ας πούμε, το πακέτο αυτό για τα αεροδρόμια. Γι' αυτό έχω στο μυαλό μου περισσότερο. Εσείς με πολύ άξινο τρόπο μας είπατε ότι... Μας είπατε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Νομίζω ότι είναι η σωστή προσέγγιση αυτή. Και εμείς ως ε, φιλελεύθεροι, μαζί με τους άλλους συναδέλφους, σας εκφράζουμε τη διάθεση για συνεργασία, ούτω ώστε να προχωρήσουμε χάρη σε αυτή τη μέθοδο και να προχωρήσουμε με αυτή τη φιλοδοξία. Καλή δουλειά, Υπουργέ. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ, για την παρουσίασή σας. Κάποια από τα θέματα που αναφέρατε θα ήθελα να τα σχολιάσω κι εγώ. Καταρχάς, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τη χρηματοδότηση. Όπως ξέρετε, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα και το αναφέρατε κι εσείς των ε, πολλών τεράστιων απαιτήσεων οικονομικών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό. Ε, τώρα έχουμε και αυτή την ε, εφεύρεση του, της διευκόλυνσης του μηχανισμού για τη χρηματοδότηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δώσουν λιγότερα χρήματα. Απλώς σημαίνει ότι ίσως να είναι λιγότερο προφανές ότι πρέπει να δώσουν αυτά τα χρήματα αλλά οι οίκοι δεν το πιστεύουν αυτό. Το έχουμε καταλάβει εν τω μεταξύ. Οπότε θα έλεγα, θα, τώρα είναι καιρός και νομίζω ότι η Δανέζικη Προεδρία μπορεί να το πράξει, να κάνουμε μία ενδιάμεση αναθεώρηση. Να μην αφήσουμε δηλαδή στην άκρη τα projects, αλλά να πούμε ότι στην παρούσα φάση πρέπει να κάνουμε ότι είναι εφικτό. Για παράδειγμα, το EMTS, ένα σημαντικό project, ε, υπάρχει, ήδη είναι στα να μπορούμε να το προχωρήσουμε λίγο παραπάνω. Ε, δηλαδή, να αφήσουμε κάποια μεγάλα πράγματα, να τα αναβάλουμε κάποια μεγάλα projects, γιατί δεν υπάρχουν ακριβώς τα οικονομικά κονδύλια, χωρίς όμως να δημιουργούμε και ψευδεστήσεις ότι θα, όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια. Ξέρουμε ότι αυτό είναι ψευδέστηση, το βλέπουμε. Βλέπουμε πώς διαχειρίζονται τα κράτη τα οικονομικά τους. Παρόλα αυτά κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό είναι λάθος. Καλύτερα να πούμε την αλήθεια παρά να λέμε ε, ψέματα στους Ευρωπαίους πολίτες, παρά να, παρά να γίνουμε αναξιόπιστοι. Δεύτερο, για το πακέτο για τα αεροδρόμια. Είπατε ότι σε ό,τι αφορά την ηχορύπανση θέλετε να προχωρήσετε. Προς τα πού θέλετε να πάτε όμως. Δηλαδή, Δεν μπορούμε εδώ να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει το δικαίωμα προσφυγής εάν μια πόλη ή περιφέρεια αποφασίσει ότι ας πούμε απογορεύει κάποιες νυχτερινές πτήσεις ή ε, περιορίζει τις ώρες εργασίας στα αεροδρόμια της και αυτό μετά μπορεί να αρθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό γιατί μιλούμε το να μπορούν δηλαδή τα κρατημέλη να αποφασίζουν. Μιλούμε για πολύ διαφορετικέ συνθήκε κατά από τι οποίε λειτουργούν συγγνώμη, τα διάφορα αεροδρόμια. Οπότε τα, τα, τι ανησυχίε και τα προβλήματα των ανθρώπων που ζουν κοντά σε αυτά τα αεροδρόμια θα πρέπει να τα, βάλουμε, να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα γιατί υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να, να, να μπορούμε να δούμε τα πράγματα κανονικά. Το να, το να μπορεί δηλαδή, το να πρέπει να μετακομίσουν οι άνθρωποι επειδή δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ από το θόρυβο, ε, δεν είναι επιλογή, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Για την ασφάλεια τώρα των αεροδρομίων, σας ε, έχετε δίκιο, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με, την, ε, με, τις, τις ε, διατάξεις ασφαλείας και κάτι να κάνουμε ως προς αυτό, να φέρουμε περισσότερη διαφάνεια, γιατί αυτό σημαίνει ότι ίσως κάποια πράγματα να πρέπει πια να διαγραφούν, γιατί μπορεί να είναι παροχημένα ή μπορεί να μην είναι αποτελεσματικά. Ουσιαστικό όμως είναι να να κρατήσουμε αυτά που λειτουργούν, να μην δημιουργούμε επιπλέον δομέ ώστε να περιπλέκουμε ακόμη περισσότερο το σύστημα. Και επίση η υπερφόρτωση των οδικών διόδων. Ε, τα φορτηγά στην μεταφορά των μετα... για την μεταφορά των αγαθών πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά σε ό,τι αφορά τις ώρες οδήγησης, τις, ε, το, πού κινούνται αυτά τα ε, φορτηγά, έτσι ώστε να μπορούμε να εποπτεύουμε λίγο την κατάσταση για να βλέπουμε και πώς, πώς κινείται τελικά, ε, πώς γίνεται η μεταφορά των αγαθών αυτών. Πρέπει λοιπόν να πούμε την αλήθεια ότι πολλά κράτη-μέλη είναι δεν δρούν έτσι όπως πρέπει, δεν λαμβάνουν τα μέτρα που πρέπει. Εσείς είσαστε διατεθειμένοι να εφαρμόσετε αυτά που έχετε ψηφίσει για τις οδικές μεταφορές. Πρέπει να προσέξουμε γιατί στον τομέα αυτό δεν πρέπει να δούμε... Ε, να, να, υπάρξει ένας φαύλος κύκλος, πρέπει να, να πατήσουμε ένα φρένο, πρέπει να φέρουμε ε, μία ισορροπία στους, ε, στις διάφορες, στα διάφορα είδη μεταφορών. Πρέπει να φέρουμε τάξη στο σύστημα γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. this... Ο τελευταίος ομιλητής, ο κ. Κόλιτσεκ από τους Γκουέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Κοιτάξτε με που είμαι. Πρώτο σημείο για τις ενέργειες μεταφορές. Πώς θα διαπραγματευτείτε με τους εταίρους για να καθοριστούν οι προϋποθέσεις για τις ενέργειες μεταφορές. Ε, ειδικά μιλάω για τα αεροδρόμια. Για να εξασφαλίσουμε το βέλτιστο ανταγωνισμό. Σημείο 2. Ποτάμιες μεταφορές. Έχετε κάποιες ιδέες πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτές τις μεταφορές, ειδικά στην ε, κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Τρίτο σημείο. Συνδεδομικές μεταφορές. Το πρώτο πακέτο. Ε, νομίζω ότι το μέλλον των συνδυοδρόμων έγκυται στη διατροπικότητα. Είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό από να κάνουμε ένα διανομή των συνοδομικών μεταφορών. Τέταρτον, οδικές μεταφορές και ασφάλεια. Το συζητήσαμε λιγάκι. Θα πρέπει να βάλουμε και την ε, κατάρτιση των ε, οδηγών. Ε, μιλάω για τα πιο αδύναμα, τους πιο αδύναμους κρίκους της αλυσίδας. Δηλαδή τους οδηγούς Πώς, έχετε κάποιες ιδέες για το πώς θα εξασφαλίσουμε τις βέλτιστες οδικές μεταφορές. Κύριε Προεδρεύοντα, θέλετε να απαντήσετε σε αυτές τις πρώτες ερωτήσεις των συντονιστών. Μετά θα μπούμε στο δεύτερο γύρο. θα μιλήσουν οι υπόλοιποι ευρωβουλευτέ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς, σας ευχαριστώ όλους για τις καλές συμβουλές που μου δώσατε. Τις οποίες θα μεταφέρω, θα επιστρέψω δηλαδή με αυτές τις συμβουλές στη Δανία. Και σας ευχαριστώ βεβαίως πολύ και για τις ευχές σας, για την Προεδρία μας. Πολύ πήραν το λόγο για συγκεκριμένα σημεία. Καταρχάς να κάνω κάποιες ε, γενικές παρατηρήσεις. Η κυρία Λίχτεμπεργκ μιλούσε για τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για να κάνουμε όλες αυτές τις αλλαγές. Φυσικά όταν μιλάμε για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, είναι σημαντικό ε, αυτά τα έργα να έχουν μια προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Μου άρεσε η παρέμβαση του Επιτρόπου σε αυτό το σημείο και τα όσα είπε για αυτό το σημείο. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει, να υπάρχει αυτά τα έργα, σε όλα αυτά τα έργα ε, ευρωπαϊκή διάσταση. Φυσικά, εγώ ως ε, Υπουργός Μεταφορών θα πρέπει να εξασφαλίσω ο πλευρά μου τους απαραίτητους πόρους και μην ξεχνάμε ότι από τη μία υπάρχει μια τεράστια κρίση στην Ευρώπη που προκάλεσε φοβερή ανεργία και από την άλλη τα μεγάλα έργα υποδομών έχουν μια, ένα δυναμικό δημιουργία θέσεων απασχόληση. Αν θέλουμε λοιπόν ανάπτυξη στην Ευρώπη, αν θέλουμε κινητικότητα στην Ευρώπη, θα πρέπει να έχουμε ένα καλό σύστημα μεταφορών, που παράλληλα δημιουργεί και θέσει απασχόληση. Αυτά τα 31,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με θετικό τρόπο. Εγώ σας το εγγυώμαι. Θα πρέπει να τα ρίξουμε στην ανάπτυξη των Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ο κύριος Γκρός έκανε συγκεκριμένα ερωτήματα για τους σιδηροδρόμους. Μίλησε για τις ρυθμιστικές αρχές στις διάφορες χώρες. Έχω την αίσθηση, αυτή τη στιγμή συζήτησα και με την ε, εισηγήτριά σας, ότι έχει γίνει ήδη σε αυτόν τον τομέα μια σημαντική πρόοδος. Και πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας θα γίνουν και άλλα πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε κοινούς κανόνες, αυτό έχω στο μυαλό μου, για τις ρυθμιστικές αρχές, με τις οποίες να λειτουργούν δηλαδή όλες οι ρυθμιστικές αρχές. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία βάση για τις, με, τις μεταφορές και για τα εμπορεύματα και για τους επιβάτες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε να κινηθούμε με περισσότερη φιλοδοξία για αυτό το πακέτο των σιδηροδρόμων. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το πακέτο αυτό. Ο κύριος Γκρός επίσης μίλησε και για τον ενιαίο ουρανό, το Single Sky. Κύριε Γκρός, συμφωνώ απόλυτα με τις προτεραιότητες που θέσατε εσείς και που έθεσε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που έχουν εντοπιστεί και από τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ συγκεκριμένα, να συνεργαστούμε. Φυσικά αυτό εξαρτάται και την καλή θέληση των κρατών μελών, αυτή η καλή συνεργασία. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με τις προτεραιότητες που αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Γκρός. Εν συνεχεία, μιλήσατε για την προσθέμενη αξία των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Νομίζω ότι σας μίλησα για τον προϋπολογισμό. Ε, σας είπα ότι θα πρέπει να έχουμε επαρκείς πόρους. Θα πρέπει να έχουμε τα λεφτά για αυτά τα έργα, προφανώς. Αλλιώς δεν θα προχωρήσουν. Το πακέτο για τα αεροδρόμια επίσης αναφέρθηκε από πάρα πολλούς. Και μιλήσατε επίσης για τα δικαιώματα των εργαζομένων στα αεροδρόμια. Αυτό είναι ένα τομέα που δεν έχω αρμοδιότητα για να σα απαντήσω. Αλλά για μένα το πρόβλημα είναι το εξή. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίε εδάφου οργανώνονται, οργανώνονται ε, με, καλύτερο τρόπο. Ε, υπέρ των εταιριών που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια, αλλά και των επιβατών που τα χρησιμοποιούν. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχουν μεγάλα κομβικά αεροδρόμια, αλλά και αεροδρόμια πιο μικρά. Και προφανώ δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα αεροδρόμια με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπαίνουν όλοι στο ίδιο καλούπι. Θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε το πακέτο ε, για τα αεροδρόμια. Θα επικεντρωθούμε στο ground handling, δηλαδή στι υπηρεσίε εδάφου, και στην ηχορύπανση. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά σημεία και νομίζω ότι μπορεί εκεί να συνεισφέρουμε. Προσπαθώ να είμαι όσο να τον πιο ακριβή στις απαντήσεις μου, να κοιτάξω λίγο τις σημειώσεις μου, με συγχωρείτε. Για τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ουρανό νομίζω ότι σας απάντησα. Τώρα. Γι' αυτό που είπαν οι φιλελεύθεροι. Σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια. Τα έργα που έχουμε προκλέψει θα προχωρήσουν. Η Δανία είναι πολύ προσεκτική γιατί θέλει η Προεδρία της να καταφέρει κάτι το οποίο θα παραδώσει στην επόμενη Προεδρία με την επο... Ε, που είναι η Κυπριακή. Ε, γι' αυτό θέλουμε στενή συνεργασία και με την προηγούμενη Προεδρία αλλά και με τη μελλοντική Προεδρία. Έχουμε την υποχρέωση να δουλέψουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι να κάτσουμε στη γωνιά μας. Ε, δεν θα προωθήσουμε τις δικές μας έτσι, εθνικές προτεραιότητες, θα έχουμε ένα όραμα πιο ευρύ, πιο ανοιχτό. Ε, και αυτή, αυτή την άποψη θα σας την πούν και όλοι οι υπόλοιποι οι Δανείοι υπουργοί. Πρέπει να κάνουμε έτσι μια δουλειά τεχνίτη, αν θέλετε. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή μηχανή που θα συνεχίσει να λειτουργεί και του επόμενου μήνε. Όχι μόνο αυτό το εξάμεινο, δεν σκεφτόμαστε μόνο αυτό το εξάμεινο. Επίση, συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε προτεραιότητε και ότι θα πρέπει να είμαστε και φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστέ. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε στόχους να υλοποιήσουμε σε καμία περίπτωση. Δεν έχει νόημα να είμαστε θεροβάμονες, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και ακριβώς έτσι πως να σας μιλήσω, με ρεαλισμό, να σας μιλήσω για στόχους που μπορούμε να υλοποιήσουμε, που μπορούμε να πετύχουμε στην Προεδρία μας. Κυρία Λίχτεμπέργκερ, σας απάντησα συμφωνώ ότι θα αναλύσουμε τα πράγματα πιο λεπτομερώς, θα δούμε τις προτεραιότητες. Φυσικά, για να δουλέψουμε καλύτερα θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πιο βιαστικές προτεραιότητες, πιο, οι πιο α, σημαντικές. Ε, ε, έγιναν ερωτήσεις για την ηχορύπανση. Δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι πολύ ακριβής ε, εδώ, αλλά το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο θόρυβος, η χορύπανση, ε, έχει επιπτώσεις ε, στους ανθρώπους καταρχάς που ζουν γύρω από τα αεροδρόμια. Πρέπει να ρυθμίσουμε διάφορα πράγματα, να έχουμε κανόνες, αλλά θα πρέπει επίσης να απαιτήσουμε από τους παραγωγούς των αεροπλάνων ε, για να κατασκευάσουν τα αεροπλάνα με ορισμένε προδιαγραφές. Υπάρχουν μια σειρά από προδιαγραφές που δεν θα πρέπει να λησμονούμε. Φυσικά θα πρέπει να δούμε και τη σχέση κόστους-οφέλους. Αυτή τη σχέση ποτέ δεν πρέπει να τη λησμονούμε. Τώρα, για τον έλεγχο στις οδικές μεταφορές. Στη Δανία. Άλλο, άλλη δουλειά κάνει ο Υπουργό Μεταφορών και άλλη δουλειά κάνει η αστυνομία που ελέγχει τις οδικές μεταφορές μαζί με τη δικαιοσύνη. Εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να υπάρχουν κανόνες και μετά θα πρέπει οι κανόνες αυτοί φυσικά να γίνονται σεβαστοί. Σε ό,τι αφορά τον τομέα των μεταφορών εν γέννη, σε ό,τι αφορά τα βαρέα οχήματα κτλ. Στην Δανία προσπαθούμε να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για αυτόν τον τομέα, τι οδικές μεταφορές. Ούτω ώστε να αποφύγουμε να καταστρέψουμε, να διασαλεύσουμε διάφορες δραστηριότητες, ε, διάφορα εμπορεύματα κτλ. Και αυτό θα είναι μια από τι προτεραιότητε τη Δανέζική Προεδρία. Ε, για το προσωπικό των αεροδρομίων νομίζω ότι απάντησα. Σε ό,τι αφορά τις ε, ποτάμιες και εσωτερικές γενικά μεταφορές, θα ήθελα να σας απαντήσει ο, ο επόμενος Υπουργός, ο Λεζόν. Θα σας μιλήσει για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές και θαλάσσιες και πλωτές εσωτερικές μεταφορές. Εγώ ως υπουργό μπορώ να σας πω πάντως ότι με μια μεγάλη προσπάθεια θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε κάποια, κάποιες από τις μεταφορές προς τις ε, πλωτές μεταφορές. Αυτή την ερώτηση όμως μπορεί να σας απαντήσει ο επόμενος υπουργό που θα μιλήσει. Προσπάθησα να απαντήσω όσο μπόρεσα σε όλες τις ερωτήσεις που μου απευθύνατε. Ευχαριστούμε, Χάρικ. Ήσουν ε, μέσα και περιεκτικός. Ε, πάμε στο δεύτερο γύρο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το φιλόδοξο πρόγραμμά σας. Είπατε βέβαια ότι πρέπει να θέσει κανείς προτεραιότητες κτλ. Αλλά στην αρχή ε, μιλήσατε για όλες τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στον τομέα των μεταφορών. Ε, μιλήσατε για την πράσινη ανάπτυξη. Νομίζω ότι οι σιδηρόδρομοι όπως και οι θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να προωθηθούν το, το καταστήσατε και εσείς αυτές, είπατε ότι ε, αυτό θα, θα, το δείτε και στην αναθεώρηση και όχι μόνο εκεί, αλλά και θα προβλέψετε κάτι για την ε, καλύτερη χρηματοδότηση των σιδηροδρόμων, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη ισορροπία για τις επενδύσεις στις διάφορες υποδομές. Λυπούμε που σε αντίθεση με αυτό, ε, για αυτά τα μεγάλα βαρέα οχήματα δεν ε, μα είπατε κάτι και για τα μεγάλα πλοία που κάνουν τι μεγάλες θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό πώς ε, μπορείτε να το ρυθμίσετε, ειδικά για τις χώρε δια, για να υπάρξει και μια, ένα αλφα επίπεδο ασφάλειας στις μεταφορές αυτές. Σκέφτεστε να προχωρήσετε αυτό το φάκελο και θα παίξετε το ρόλο του ενδιάμεσου, τι ακριβώ σκέφτεστε να κάνετε. Επίση, το θέμα τη ασφάλεια των οδικών μεταφορών είναι ένα σημαντικό θέμα και επίση οι κοινωνικέ διατάξει. Η κοινωνική πτυχή είναι ένα θέμα, αλλά η ασφάλεια και οι κυρώσει στις φυσιολογική, δηλαδή στις φυσιολογικές οδικές μεταφορές, όχι για, όχι για τα μεγάλα βαρέα οχήματα ή τα φορτηγά, ε, πώς, πώς, θα το, πώς, θα, πώς θα το ρυθμίσετε να υπάρξουν, να υπάρξουν και κάποιες ποινικές σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή οτιδήποτε. εδώ υπάρχει και μια ρήτρα opt-out. Σκέφτεστε παρόλα αυτά να συμβάλλετε για αυτή την διασυνοριακή συνεργασία για τον τομέα αυτό της ασφάλειας. Γιατί νομίζω ότι και η κατάρτιση, η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση είναι πολύ σημαντική τομή. Αλλά χωρί κυρώσει στι οδικέ μεταφορέ δεν θα επιδευθεί ο στόχο μα. Ευχαριστώ. Κύριε Σαναλόβα. Ευχαριστώ. Ούτε κι εγώ έχω διερμηνία στη γλώσσα μου. Θα επιχειρήσω να μιλήσω στα αγγλικά. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίαση των στόχων και του προγράμματος της Δανικής Προεδρίας. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι που δεν επισημάνατε ρητά στις προτεραιότητες, στο θέμα της οδικής ασφάλειας, που ήδη ανέφεραν οι προλαλήσαντες. Εμένα με ενδιαφέρει κυρίως η πανευρωπαϊκή ε, εφαρμογή του αυτόματου συστήματος ε, συναγερμού για την οδική ασφάλεια. Ποια είναι η θέση της δανικής κυβέρνησης για τον ηλεκτρονικό αυτό κώδικα, ευρωπαϊκό κώδικα και είπατε ότι ε, η οδική ασφάλεια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το περιβάλλον. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για τα εξαιρετικά αγγλικά σας. Ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω κάτι γι' αυτό. Μας δώσατε ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι με το πρόγραμμα και στη σελίδα 7 λέτε ότι θέλετε να συνεχίσετε τον αγώνα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τι ε, μεταφορές γιατί αυτές οφείλονται, ε, σε αυτές οφείλεται το 30% των ε, εκπομπών αερίων. Και ε, από αυτό το 30% το 80% ανήκει στις ε, οδικές μεταφορές. Και εκεί μιλάμε για τα τεράστια αυτά φορτηγά που ε, μολύνουν την ατμόσφαιρα. Ξέρετε το πρόβλημα που υπάρχει στην Γερμανία. το, η, το, η κάτω βουλή ήθελε να, το, να μην το περάσει από την πάνω βουλή. Ξέρουμε ότι γίνεται μία μελέτη η οποία λέει ότι ε, το 38% των ε, μεταφορών θα πάει από τις οδικές μεταφορές στους ε, σιδηροδρόμους. Αν δηλαδή θέλετε να ενισχύσετε, τις, τους, αν θέλετε να αυξήσετε τις εκπομπές στις οδικές μεταφορές και να ενισχύσετε τις οδικές μεταφορές, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε ακριβώ αυτά τα τεράστια φορτηγά να κάνουν τι μεταφορέ. Πρέπει το, να υπάρξει κοινωνική πτυχή σε όλη αυτή την ε, ε, κατανομή του κόστου. Υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και το κέρδο πάντα καταλήγει τελικά στα χέρια λίγων. Πρέπει να υπάρχουν όμω ε, κοινωνικά κριτήρια εδώ. Αν πείτε εσεί ότι πρέπει να πληρώσετε για τι υποδομέ, ε, κανένα δεν θα ζητήσει να ε, βάλει αυτή, αυτά τα τεράστια φορτηγά στου δρόμου, γιατί προφανώ κοστίζουν πάρα πολύ. Μετά. Ξαφνικά το τούνελ είναι πολύ πιο φτηνό ε, το να περάσει κανείς ε, από ότι ε, η Γερμανία. Ξέρετε ότι η Δανία πλήρωσε την γέφυρα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες μας γιατί η Γερμανία δεν το ήθελε. Οπότε όταν κάποιος πληρώνει μπορεί να πει και όχι. Αλλά η Γερμανία υποσχέθηκε ότι θα συμβάλλει. Κανεί δεν ξέρει από πού θα προκύψουν αυτά τα λεφτά γιατί είναι πάρα πολλά. Δεν μιλάω ούτε για την Ιταλία ούτε για τη Γερμανία. Μιλάω για 14 συμβάσει διασυνοριακέ, τι οποίε μέχρι τώρα η Γερμανία δεν έχει, α, δεν έχει ε, τηρήσει. Δύο έχει τηρήσει μόνο από αυτέ τι 14 που έχει υπογράψει. Τι 12 τι έχει παραβιάσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό τον προς πίσω δεν βοηθάει. Οπότε καλύτερα θα ήταν να εξηγιάνετε του σιδηροδρόμους για να μπορεί κανείς να πάει από το ρώστο ας πούμε στο Βερολίνο και θα έχετε κι εσείς πολύ λιγότερα προβλήματα από την Κοπενχάγη. Επίσης, αναθεώρηση, αναδιατύπωση, η ρύθμιση ναι είναι σημαντική, κάναμε ήδη τη συζήτηση. Εσείς θέλετε να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο αυτά τα, θα δίνονται οι άδειε ή δεν θα δίνονται. Αν ναι, τότε πείτε μας. Μέσα σε ένα μήνα θα γίνεται αυτό. Αλλά όταν έχει συμπληρωθεί σωστά το έντυπο. Ε, γιατί ποτέ τα κρατη μέχρι τώρα δεν είχαν συμπληρώσει σωστά τα έντυπά του. Πείτε ότι θέλουμε σε ένα μήνα να γίνει αυτό. Αν, ένα, αν δεν έχει συμπληρωθεί, ο, αν έχει συμπληρωθεί ο ένα μήνα, πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε γίνεται, συμπληρώνεται η αίτηση. Αν συμπληρώνεται, στείλτε τη. Αν δεν τη συμπληρώνεται, ακυρώνεται η άδεια. Χρειαζόμαστε σαφεί κανόνε, χρειαζόμαστε σαφεί αποφάσει, δεν χρειαζόμαστε άλλο μπρο πίσω και άλλη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την ενημέρωση. Ε, όπως ε, νομίζω προκύπτει από τη συζήτησή μας για τον φάκελο των μεταφορών, το 2012 είναι έτος των διευρωπαϊκών δικτύων. Γνωρίζετε ότι η επόμενη αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών έχει προβλεφθεί για, για το 2023. Επομένως δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα διαμορφώνουν την εικόνα της Ευρώπης του μέλλοντος το ότι βρισκόμαστε, κύριε Υπουργέ, αντιμέτωποι με την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες της, δεν πρέπει να είναι αιτία ή αφορμή να καθυστερήσουμε. Αντιθέτως πρέπει να είναι κίνητρο για να επιταχυνθεί η διαδικασία προετοιμασία αυτού του μεγάλου project των διευρωπαϊκών δικτύων. Ε, η Ευρώπη, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, έχει ανάγκη από μια ευρωπαϊκή επιτυχία. Και νομίζω ότι ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα δίνουν αυτή την δυνατότητα. Επομένως, καλείστε ως Προεδρία να διασφαλίσετε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αυτού του μεγάλου project, αναπτυξιακού project. Θα πρέπει να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, να τα αντιμετωπίσουν και εκείνα ως ευρωπαϊκό project και όχι να έρθουν με αποσπασματικές, αμυγός και αποκλειστικά εθνικές προτεραιότητες, κάτι που θα καθυστερήσει την προσπάθεια για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας πρέπει στη συγκεκριμένη ειδικά περίπτωση να είναι κυρίαρχος και όχι οι εθνικές προτεραιότητες. Ε, και βεβαίως περιμένουμε να δούμε την Προεδρία να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις ευαισθησίες, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του Κοινοβουλίου, ειδικά σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα δύο θέματα, αν μπορέσετε συγκεκριμένα να μου δώσετε έστω μια γρήγορη απάντηση. Πώς αντιμετωπίζει η Προεδρία το θέμα των προδιαγραφών για τις υποδομές στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων και πώς το θέμα των διαδρόμων. Ε, αν μπορείτε με μία σύντομη απάντηση για να έχουμε ήδη από τώρα μια εικόνα ποιε είναι οι σκέψεις της Προεδρίας πάνω σε αυτά τα δύο ζητήματα. Και ένα τελευταίο, δεν θέλω βεβαίως να επιβαρύνω μια ήδη πολύ φιλόδοξη ατζέντα που έχετε, αλλά κύριε Υπουργέ δεν ακούσαμε κάτι για το φλέγον ζήτημα της αντιμετώπισης της πειρατείας που γνωρίζω ότι είναι ένα από τα θέματα προτεραιότητος και ειδικού ενδιαφέροντος για τη Δανία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Mr. Ευχαριστώ κύριε Φιντάντσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλή τύχη και πολλές ευχές ε, Υπουργέ. Πάρα πολλά έχουν υποθεί ήδη, αλλά πολύ γρήγορα θέλω να πω και εγώ για το πακέτο για τα αεροδρόμια. Πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε την ε, τύχη και την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για τις προτάσεις της Κομισιόν, για τις ονοβυρίδες ας πούμε. Ε, πώς μπορούμε, χρησιμοποιώντας καλύτερα τα σλότ, να αυξήσουμε το δυναμικό και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα αεροδρομιά μας. Ε, επίσης, για το ground handling, για τις υπηρεσίε εδάφους, ε, αν μπορούμε να έχουμε καλύτερες δράσεις, ούτως ώστε να αυξήσουμε, να ανεβάσουμε τα πρότυπα παροχής ε, υπηρεσιών μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε για την τεχνολογία RTMS. Ε Πιστεύω ότι είναι θέμα προτεραιότητας. Ξέρω ότι μια χώρα όπως η δική σας έχει επενδύσει πάρα πολύ για να αυξήσει την ασφάλεια. Πιστεύω ότι αυτή μπορεί να είναι μια καλή πρακτική που μπορούμε να την εξάγουμε ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να επανέλθουμε λίγο στον ενιαίο ουρανό. Υπενθυμίσατε πολύ σωστά, ή μάλλον ο ο συντονιστή μου, ο κύριο Γκρό, μίλησε για τα FAB, για τα FABs. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, εξίσου σημαντικό, το ΣΕΖΑΡ, για τη διαχείριση τη ε, εναέρεια κυκλοφορία. Είμαστε στην τέταρτη φάση εφαρμογή αυτού του προγράμματο αυτού του έργου. Ε, και οι ιδιωτικέ εταιρείε, αεροδρόμια, αεροπορικέ εταιρείε, διαχειριστέ τη εναέρεια κυκλοφορία έχουν επενδύσει πάρα πολύ, έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ. Υπάρχει επίση μια δέσμευση από τα κράτη-μέλη να βάλουν τρία από τα 30 δι για την υλοποίηση αυτή τη ε, φάση, που είναι τρίτη, συγγνώμη, όχι τέταρτη. Αλλά όμω ε, δεν το αναφέρατε ω προτεραιότητα αυτού του έξι μήνε προεδρίας σα. Πιστεύω όμω ότι μπορείτε να δουλέψετε και αυτού του έξι μήνε μαζί με την ε, Κυπριακή Προεδρία που θα σα ακολουθήσει, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε αυτά τα τρία δι, ε, τρία από τα 30, έτσι ε, είναι σημαντικό αυτό το ποσό γιατί αν ξεκινήσουμε τα τρία μπορεί να βρούμε και τα υπόλοιπα 27 για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ. Ευχαριστώ. Καντσιάν, τελευταίος αλλά σημαντικός. Ευχαριστώ και πολλές ευχές Υπουργέ. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο, μόλις τώρα και ο Σφιντάντσα. Μαζί με αυτά τα λεφτά που θα βάλουν τα κράτη-μέλη, Μπορούμε να προωθήσουμε το ΣΕΖΑΡ. Αλλά επίσης μην ξεχνάμε και το GMS, GMES, το οποίο το έχουμε ξεχάσει στον προϋπολογισμό. Αυτή την συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού τομέα για να προωθήσουμε αυτά τα έργα. Τώρα, κάτι πιο γενικό, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των υποδομών, κύριε Υπουργέ. Εμείς Σήμερα έχουμε ε, μιλάμε για αυτά τα 31,7 δις. Αν δεν τα ξοδέψουμε, αν δεν τα δώσουμε ως επιδοτήσεις, ας πούμε, όπως έγινε στο παρελθόν, μπορούμε να προωθήσουμε κάποια έργα υποδομών. Δεν πιστεύετε ότι ένα τμήμα αυτών των ε, χρημάτων θα μπορούσε να προέλθει από το ταμείο που έχει προβλεφθεί, το ad hoc ταμείο. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τα διάφορα ταμιευτήρια των κρατών μελών δεν θα, μπορούν, δεν θα μπορούσαν να συνεργαστούν ούτως ώστε να φτιάξουν ένα ad hoc ταμείο όπως κάναμε για την ενέργεια. Ίσως σε μικρότερο βαθμό. Για να εξασφαλίσουμε, το κάναμε για να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο σημαντικό ταμείο για να βοηθήσουμε ε, την υλοποίηση αυτών των μεγάλων έργων υποδομών. Αυτή την ερώτηση την κάναμε πρώτη φορά ε, εδώ και δυόμιση χρόνια και την επαναλαμβάνουμε κάθε τόσο στην, ε, στις ε, διάφορες προεδρίες. Κάθε φορά μας λένε ναι. Αλλά τουλάχιστον εσείς προσπαθήστε, προσπαθήστε. Αυτά τα 31,7 δις, από αυτά μάλλον, ένα τμήμα να το βρούμε μέσα από το, τους τρόπους που σας είπα. Επίσης, τα ευρωομόλογα. Χάρη σε αυτά θα μπορούσε να χρεωθεί η Ευρώπη, θα μπορούσε να δανειστεί δηλαδή, για να χρηματοδοτήσει κάποια πράγματα. Για να υλοποιήσει κάποια έργα. Νομίζω ότι για να υλοποιήσουμε αυτές τις μεταφορές θα πρέπει να κάνουμε τέτοιου τύπου προσπάθειες. Επίσης μην ξεχνάτε Υπουργέ ότι το να βιαστούμε είναι σημαντικό γιατί πιέζει ο χρόνος. Τώρα για τα δικαιώματα των επιβατών. Δεν άκουσα να λέτε τίποτα. Θα θέλαμε να σας ακούγαμε, να λέτε κάτι για τους επιβάτες θα θέλαμε ε, να υπάρχουν παντού τα ίδια δικαιώματα για τους επιβάτες, για όλα τα μέσα μεταφορών. Ε, υπάρχει κάτι σχετικό στο πρόγραμμά σας για τους 6 μήνες για τα δικαιώματα των επιβατών. Ευχαριστώ. Κύριε Προεδρεύοντα, έχετε το λόγο. Θα ξεκινήσω με την τελευταία παρατήρηση του κυρίου Καντσάν. Δεν πολύ κατάλαβα την τελευταία σας ερώτηση. Δηλαδή, εμείς θα πρέπει να εγγυηθούμε για τα δικαιώματα όλων των επιβατών α, α, ανα πάσα περίπτωση, δεν νομίζω. Ε, παρά είναι μεγάλο, μεγάλη ευθύνη για ένα και μόνο άνθρωπο. Σίγουρα η πολιτική των καταναλωτών μας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των επιβατών. Γιατί οι επιβάτε είναι και αυτοί πελάτες, καταναλωτέ. και σίγουρα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα δικαιώματά σου, αλλά το να εγγυηθούμε τα πάντα σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω. Κύριε Καντσάν, αναφέρθηκε και μία άλλη χρηματοδότηση και αυτό είναι το θέμα της διάσκεψης της Κοπενχάγης υπάρχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης για να ε, χρηματοδοτήσουμε μεγαλεπίβολα σχέδια. Μιλούμε για συμπράξεις ε, δημοσίου ε, και ιδιωτικού, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ελάχιστα κρατικά κονδύλια, γι' αυτό θα πρέπει να αναζητήσουμε και εναλλακτική χρηματοδότηση και να αξιοποιήσουμε φυσικά το στο έπακρο τα κονδύλια που διαθέτουμε. Σε αυτή τη διάσκεψη λοιπόν θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βρούμε κονδύλια εκεί που έχουμε ελλείψεις. Και μία απάντηση γενική που καλύπτει την ερώτηση ε, ορισμένων συναδέλφων για τα φορτηγά μεγαθύρια, για αυτές τις τεράστιες νταλίκες. Ακόμη και οι φιλοπεριβαλλοντικές οικολογικές οργανώσεις στη Δανία έδειξαν ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και ευωδόθηκαν πολλές πρωτοβουλίες για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να αποδείξουμε ότι εμπορεύματα που μεταφέρονται με τέτοιου είδους μεγαθύρια φορτηγά, τέτοιου είδους μεταφορές έχουν ε, θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και για το κλίμα. Σίγουρα θα πρέπει να μεταφερθούν τα εμπορέματα από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β και με λογικό τρόπο. Αυτά όμω τα μεγαθύρια φορτηγά αυτέ ε, ε, οι ε, δεν χρειάζεται να καλύπτονται από νέε διατάξει. Αν δύο χώρε έχουν δεχθεί την κυκλοφορία στο έδαφος τους αυτών των μεγάλων φορτηγών, αυτών των Ιταλικών, γιατί να μην μπορούν να το συμφωνήσουν, άμα δύο χώρες επιθυμούν να το επιτρέψουν. Νομίζω ότι είναι λογικό, εφόσον συμφωνούν οι χώρες ε, να κυκλοφορούν τέτοια μεγαθύρια φορτηγά στους δρόμους τους, ε, να είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Μιλήσαμε και για την πράσινη ανάπτυξη, τη φιλοπεριβαλλοντική ανάπτυξη. Ε, έχει κάποια σχέση και με αυτά τα μεγάλα φορτηγά. Νομίζω όμως ότι σε τέτοιου είδους συζητήσεις θα πρέπει να πριτανεύει η λογική, ο κοινό νου και ο ρεαλισμό. Δεν, χρειάζεται, δεν χρειάζονται κατά ανάγκη νέε διατάξει, αρκεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ δύο χωρών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στη Δανία, έχουμε πολλέ επιτροπέ ε, που κάθε μία είναι καθήλια αρμόδια για άλλο τομέα. Και μερικέ φορέ ε, ορισμένα ντοσιέ εμπίπτουν σε αρμοδιότητες ε, περισσότερων επιτροπών. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας και στην Κοπεχάγη και εδώ θα δώσουμε την έμφαση στην ασφάλεια των νέων, των παιδιών και γι' αυτό θα οργανώσουμε και σχετική διάσκεψη για την ασφάλεια των παιδιών και των νέων. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησε σε ερωτήσεις κυρία Σενάλοβα ε, νομίζω και στις ερωτήσεις του κυρίου Κράμερ για αυτά τα τεράστια φορτηγά. Και δύο παρατηρήσεις για την ε, συνδεση δενιας Δανίας-Γερμανίας. Εγώ μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχα ασχοληθεί με το σημείο αυτό, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις γερμανικές αρχές. Και όταν η Δανία και η Γερμανία συνάπτουν μια συμφωνία και οι δύο χώρες τηρούν τους όρους αυτής της συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών, και εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να δρούμε λαμβάνοντας υπόψη και το περιβάλλον και το κλίμα. Και γι' αυτό και η σύνδεση ε, Δανίας-Γερμανίας και από περιβαλλοντική άποψη είναι σημαντική τα εμπορεύματα από τις σκανδιναβικές χώρες ε, με προορισμό την ε, κεντρική Ευρώπη σήμερα κυκλοφορούν με διαφορετικό τρόπο χάρη, σε αυτούς τους διαδρόμους, χάρη σε αυτές τις γέφυρες και τις διασυνδέσεις. Και παρόλο που δεν συμφωνούμε απόλυτα μεταξύ μας, θεωρώ ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα και για το κλίμα και για τις μεταφορές των εμπορευμάτων. Τέθηκαν πολλές εύστοχες ερωτήσεις Προσπαθώ εδώ να τις κατατάξω ανάλογα με το θέμα τους. Κάποιος μίλησε για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και συμφωνώ με αυτά που είπατε ότι θα πρέπει να περιέχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να μην χρηματοδοτούν μόνο τοπικά και περιφερειακά σχέδια δεν αρκεί ο τοπικός και περιφερειακός χαρακτήρας. Θα πρέπει ε, να είναι αποδοτικές αυτές οι επενδύσεις και να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση. Φυσικά θα πρέπει και οι χώρες να συμβάλλουν στην δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για να δημιουργηθούν αυτοί οι ευρωπαϊκοί διάδρομοι. Αυτή την άποψη λοιπόν όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν και σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όταν θα ολοκληρώσουμε αυτούς τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα προστιθέμενη αξία. Σε ό,τι αφορά την πειρατεία, όντως η πειρατεία είναι οξύδωτο πρόβλημα, αλλά παραπέμπω το ζήτημα στο συνάδελφο, τον Λεσόλ, που είναι αρμόδιος για τις θαλάσσιες μεταφορές και θα θίξει το θέμα αυτό στη δική του παρέμβαση. Ο κύριος Φιντάντσα Ζητώ συγγνώμη κύριε Φιντάντσα αν δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Κύριε Φιντάντσα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι χρειαζόμαστε κάποιες ε, θεμελιώδεις ενέργειες. Αυτές οι βασικές ενέργειες είναι σημαντικές και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτές. Όταν μιλούμε για το πακέτο για τα αεροδρόμια, έχουμε τις ε, δράσεις ε, για τις υπηρεσίες εδάφους και τα μέτρα για τον περιορισμό του θορύβου. Η Ιδανική Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει το ντοσχέ αυτό, αλλά το ζητούμενο να καθορίσουμε κάποιες προτεραιότητες. Αποφασίσαμε στη Δανία να επικεντρωθούμε στη, στο έδαφος. Αυτό δεν σημαίνει θα αδρανίσουμε στους, επόμενους, στους υπόλοιπους τομείς, αλλά θα επικεντρωθούμε κυρίως στις υπηρεσίες εδάφους. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Αν παρέλειψα ορισμένες, ε, μπορούμε στη συνέχεια να τις απαντήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Πραγματικά προσβλέπουμε στην συνεργασία μας μαζί σας κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε στο τέλος του εξαμήνου για να μας κάνετε μια αναφορά για το πώς προχωρήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς ε, και τους συναδέλφους σας που ήσασταν σήμερα εδώ και βεβαίω ε, ισχύει πάντα η πρόσκλησή μα ε, να έρχεστε εδώ. Βεβαίω εμεί πάντα είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και την Προεδρία του για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Κάποιε φορέ, ε, τα θαύματα αργούν λίγο να γίνουν, κάποιε άλλε η συνεργασία βοηθάει. Οπότε η δική μου πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Είμαι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Συνάδελφοι, μια μικρή διακοπή για να αλλάξουμε υπουργού. Δεν εννοώ ανασχηματισμό κυβέρνηση φυσικά. Απλώς περιμένουμε τον ε, επόμενο υπουργό, τον κύριο Σον, που θα μας αναπτύξει το θαλάσσιο σκέλος της Δανικής Προεδρίας. Okay, Πάμε στο επόμενο σημείο, ανταλλαγή απόψεων, με τον Δανό Προεδρεύοντα, που είναι Υπουργό ε, Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης, ο ΣΟΝ αλλά είναι και υπεύθυνο ταυτόχρονα με τις θαλάσσιες, για τις θαλάσσιες μεταφορές. Κύριε Υπουργέ, Έχουμε διάφορους φακέλους ανοιχτούς για τις θαλάσσιες μεταφορές και ελπίζουμε να τους κλείσουμε κατά τη διάρκεια της ε, ε, Προεδρίας. Ε, ελάχιστη κατάρτιση για τους ναυτικούς, ε, ο καονισμός για την ΕΦΣΑ και ε, η αναδιατύπωση του καονισμού για τα δεξαμενόπλια με διπλό κήτος. Σήμερα το πρωί ο Επίτροπος Κάλλας μας ενημέρωσε για το τι συνέβη τι συμβαίνει τώρα μετά το ατύχημα του Κώστα Κονκόρδια ε, στα νυχτά των ακτών της ε, Τοσκάνης, της Ιταλίας. Μας ενημέρωσε λοιπόν για το θέμα αυτό του Κρουαζιερόπουλου. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πείτε. Και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, σας δίνω τον λόγο κύριε Υπουργέ. έχετε το κόκκινο κουμπάκι για να ανοίξετε το μικρόφωνο σα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου στείλατε για να σας συναντήσω εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Ε, με μεγάλη χαρά έρχομαι για να συζητήσω τις προτεραιότητες της Δανέζικης Προεδρίας στον τομέα αυτό. Πριν ξεκινήσω την παρέμβασή μου, θα ήθελα εκ μέρους της Προεδρίας ως ε, υπουργό υπεύθυνο για τις θαλάσσιες μεταφορές να εκφράσω την βαθύτατη θλίψη που νιώθω για τα θύματα και τις οικογένειές τους που υπήρξαν θύματα ε, από την ε, βήθηση του Κώστα Κονκόρδια στις 13 Ιανουαρίου. Η Προεδρία θα παρακολουθήσει και τις εξελίξεις αλλά και την έρευνα που, είναι, που τρέχει αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Brian Simpson για την επανεκλογή του στην Επιτροπή Μεταφορών και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη θαυμάσια συνεργασία που πάντα είχαμε. Ε, βλέπω ότι πολλά από τα μέλη της Επιτροπής ε, παρέμειναν, παραμένουν σε αυτή την Επιτροπή, δεν άλλαξαν και χαίρομαι που θα τους ξαναδώ, που θα συνεχίσουμε τη συνεργασία. Ε, χαίρομαι που βλέπω και νέα μέλη όμως, ε, με, τους οποίους, με τα οποία επίσης θα συνεργαστώ. Το Νοέμβριο είχαμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε τους ε, συντονιστές της Επιτροπής που μου έδωσαν το πλαίσιο ε, των εργασιών στην Επιτροπή σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας εταίρος πάρα πολύ σημαντικός για την Προεδρία μας και η στόχη μας είναι κοινή, η δουλειά που κάνουμε είναι κοινή. Πρέπει να δημιουργήσουμε και αποτελέσματα υπέρ των ε, πολιτών και των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτεραιότητε είναι ο συνεχή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βέβαια, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάρουμε μαζί τι σωστέ αποφάσει, ούτω ώστε να βάλουμε στο σωστό δρόμο ε, την προσπάθεια για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ και την Πολωνική Προεδρία και την Κομισιόν για τα καλά αποτελέσματα που πετύχαμε σε θέματα πολύ σημαντικά και που πετύχαμε, τα πετύχαμε κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας και περιμένω ε, με ενδιαφέρον να συνεργαστούμε μαζί. Η Δανία πήρε την σκητάλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή πολύ δύσκολη λόγω της οικονομικής κρίσης. Ε, αντιμετωπίζουμε ίσως τις πιο έντονες ε, προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ποτέ η απόφαση να ενισχύσουμε την ε, οικονομική και χρηματοπιστωτική συνεργασία στην Ευρώπη ε, και να υπάρξει μια οικονομική πολιτική στην Ευρώπη, αυτό είναι το φλέγον θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η Δανέζικη Προεδρία θα προσπαθήσει να πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, ούτω ώστε να ενισχύσουμε, ελπίζουμε τουλάχιστον την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δείξουμε να δείξουμε την σημασία που έχει η συνεργασία στην Ευρώπη. Θα δουλέψουμε για μια Ευρώπη υπεύθυνη, δυναμική, πράσινη και ασφαλή. Είμαι πεπισμένος ότι η ανάπτυξη και η οικονομική ενοποίηση, ενίσχυση αν θέλετε, είναι δύο, τα δύο πόδια πάνω στα οποία θα πρέπει να πατήσει η Ευρώπη για να βγει από την κρίση. Και ελπίζω να, συνεργαστούμε, να συνεργαστούμε για τον κοινό μας στόχο που είναι η ανάπτυξη στην Ευρώπη. Στην Δανία είμαι υπουργό Οικονομικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης και εδώ συμπεριλαμβάνεται και η ναυσιπλοεία, οι θαλάσσιε μεταφορέ. Πρόκειται για μια οικονομική δραστηριότητα πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή οικονομία. Στο θαλάσσιο τομέα δεσμευόμαστε, ούτω ώστε η ναυσιπλοεία στην Ευρώπη να γίνει πιο ασφαλή. Και είδαμε ότι το ατύχημα του Κώστα Κονκόρδια δείχνει πόσο είναι σημαντικό να αξιολογούμε συνέχεια την, τα πρότυπα ασφάλειας που έχουμε. Θα δούμε τι θα προκύψει από την ε, έρευνα, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και τα πορίσματα της έρευνας και τα μαθήματα που θα προκύψουν από αυτό το ατύχημα και τα έρευνα θα επηρεάσουν και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εν ώψη της ε, αναθεώρησης οδηγίας για τα επιβατηγά πλοία. Ε, εμείς θα παρακολουθήσουμε πλευράς Δανέζικης Προεδρίας το φάκελο αυτό με πολύ προσεκτική ματιά. Θα δεσμευτούμε ούτως ώστε θαλάσσιες μεταφορές και η ναυσιπλοεία να γίνουν πιο πράσινες επίσης. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα επίσης του τομέα στην παγκόσμια σκηνή. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε ε, στους ναυτικούς, ε, στο πλήρωμα και στη μείωση του κόστους για τη βιομηχανία, αλλά και για τους επιβάτες. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να προωθήσουμε τους φακέλους που έχουν ήδη ξεκινήσει και που είναι επιτάπητος. Ε, ούτως ή άλλως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό του οργανισμού ΕΜΣΑ. Έχουμε τον κανονισμό ε, για τα δεξαμενόπλια διπλού κήτους. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Σε ό,τι αφορά την οδηγία STCW, ε, έχουν εγκριθεί κάποιες τροπολογίες που αναφέρθηκαν πρώτα στην... συμφωνήθηκαν καταρχήν στη Μανίλα. Θα πρέπει να έχουμε σωστά πρότυπα για, τα, για την κατάρτιση των ναυτικών, και η οδηγία μπορεί να βελτιώσει την, και την ασφάλεια στα πλοία. Το Δεκέμβριο του 2011 η Επιπολωνικής Προεδρίας ε, επιτεύχθη συνένεση στο Συμβούλιο, συμφωνία στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο ε, επικεντρώθηκε στην τροποποίηση της οδηγίας ούτως ώστε να προσαρμοστεί σε όλες τις αλλαγές, σε όλες τις ε, τροπολογίες που είχαν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι η οδηγία προσαρμόζεται ουσιαστικά ε, στα διεθνή πρότυπα. Είναι σημαντικό να καθιερώσουμε ενιαίους κανόνες προς όφελος της ναυσιπλοείας ε, και προς όφελος των ναυτικών ανά τον κόσμο. Επίσης, είναι σημαντικό για τις θαλάσσιες ε, μεταφορές να υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες παντού. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το πλήρωμα, ας πούμε, το προσλάβαμε στην Ευρώπη ή στην Ασία. Θα πρέπει να υπάρχουν τα ίδια πρότυπα. Αυτά τα συζήτησα με τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής και με τον, ε, που είναι και εισηγητής της πρότασης, που είναι ο κ. Σίμψον. Και ο κ. Σίμψον πιστεύει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό αυτοί οι κανόνες. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που θα υπάρξει αυτή η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτό το θέμα και ελπίζω ε, να προχωρήσουμε το θέμα στα πλαίσια της Προεδρίας μας. Επίσης, Περιμένουμε την πρόταση της ε, Κομισιόν για τη σύμβαση για τις ε, συνθήκες εργασίας των ε, ναυτικών. Μια άλλη πρόταση πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την, τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών είναι αυτή η οδηγία και στόχος της είναι η εναρμόνιση ούτω ώστε τα κράτη της σημαία να σεβαστούν όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν διεθνείς και ευρωπαϊκές, για τις συνθήκες εργασίας. Περιμένουμε το κείμενο της Κομισιόν. Ε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να μπορέσουμε ακόμα επί Δανέζικης Προεδρία να το συζητήσουμε. Τώρα, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στην Αυσιπλοεία, ε, είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία, ένα σημαντικός οργανισμός για την καταπολέμηση της μόλυνσης και την ασφάλεια στη θάλασσα. Ο οργανισμός αυτός θα πρέπει να συνεχίσει να είναι ένα σημαντικό φορέας. Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει ο ΕΜΣΑ να γίνει ένας ε, κεντρικός οργανισμός ε, με πολλές αρμοδιότητες και νομίζω ότι υπάρχει συνένεση γύρω από αυτή τη φιλόδοξη πρόταση. Έγινε μια συζήτηση στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, του Δεκέμβριου του 2011, και από τη συζήτηση αυτή προέκυψε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει μια πιο δυνατή έμσα, ένα πιο δυνατό οργανισμό. Επίσης, ε, θα να ευχαριστήσω τον κύριο Φλάνκεστάιν που ήταν εισηγητής αυτής της πρότασης και ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ σε με αυτό το κείμενο. Ε, και χαίρομαι και πιστεύω θα συνεχιστεί η συνεργασία μαζί του. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού ΕΜΣΑ, το, τον Ιούνιο του 2011 το Συμβούλιο κατέληξε σε κοινή θέση. Για το Συμβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό το χαρτοφυλάκιο των αρμοδιοτήτων της ΕΜΣΑ να διευρυνθεί σε τομείς όπου πραγματικά μπορεί να δημιουργηθεί προσθέμενη αξία. Και για ζητήματα που δεν μπορούν τα κράτη να δράσουν με καλύτερο τρόπο από το ευρωπαϊκό επίπεδο, άρα ο ΕΜΣΑ. Φυσικά, ε, ο ΕΜΣΑ θα πρέπει να ασχολείται μόνο τα θέματα της αρμοδιότητάς του θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους ε, δεινούς και χαλεπούς οικονομικούς καιρούς οποίους ε, περνάμε. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ε, ισορροπία μεταξύ καθηκόντων και πόρων της ΕΜΣΑ. Θα πρέπει η ΕΜΣΑ να ασχολείται με τρόπο έτσι πολύ στεναρός ότι αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα, την καταπολέμηση της ρήπανσης, αλλά μην ξεχνάτε ότι η εποχή, οι εποχές είναι χαλεπές και ζούμε σε συνθήκες λιτότητας. Επί κάποιων σημείων της πρότασης υπάρχει, υπάρχει διαφορά όμως ανάμεσα στις θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ε, γι' αυτό καλό είναι να έχουμε όλοι μας διάθεση για διαπραγμάτευση και έτσι, συνεργασία αν θέλουμε να φτάσουμε στη συμφωνία. Πιστεύω, νομίζω ότι μπορώ να πω, ότι και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πιστεύουν ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα και αξίζει να γίνει μια προσπάθεια για συμβιβασμό το Συμβούλιο έχει εκπονήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για τις επόμενες διαπραγματεύσεις και περιμένω με ανησυχία τι θα προκύψει. Ελπίζω να συνεργαστούμε, ελπίζω να υπάρξει αμοιβαία βοήθεια για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για την ε, εισαγωγή ε, δεξαμενόπλων διπλού κήτους, ε, υπάρχει σημαντική πρόοδος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτό τον κύριο Ρίλκε, τον εισηγητή, για τη δουλειά που έκανε επί του φακέλου αυτού. Τώρα, πρόκειται για μια τεχνική τροποποίηση, για μια κωδικοποίηση του καονισμού. Το Δεκέμβριο το Συμβούλιο κατέληξε συμφωνία και τώρα η Δανέζικη Προεδρία θα προσπαθήσει να πετύχει την συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ούτω ώστε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα και να υπάρξουν αυτοί οι κανόνε. Ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι αυτό της πειρατεία. Είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό για, την, διεθνή, για τις θαλάσσιες μεταφορές και ιδίω και για τους ναυτικούς που αποτελούν πλήρωμα. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βαντάλεν και τον κύριο Κουμουτσάκο για την πρωτοβουλία τους Μάλιστα, οργανώθηκε μία ακρόαση το φθινόπωρο για την πειρατεία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ήταν πάρα πολύ σημαντική, με σημαντικό αντίκτυπο. Ε, εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι η πειρατεία είναι πολύ σημαντική για την οικονομική μα δραστηριότητα και για του ναυτικού. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτό το θέμα και να το έχουμε στην ημερήσια διάταξή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή οργάνωσε προβλέπει μάλλον μια διάσκεψη 28-29 ε, Μαρτίου σε συνεργασία με τη Δανέζικη Προεδρία. Μια διάσκεψη ακριβώς για το θέμα της πειρατείας. Το, το πρόβλημα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών ε, και της πειρατείας φυσικά δεν μπορούν να επιληθούν με μία διάσκεψη που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να συνεισφέρει αυτή η διάσκεψη. Ε, μπορεί να διατηρήσει το ενδιαφέρον σε αυτό το θέμα και να σκεφτούμε τις διάφορες λύσεις. Νομίζω ότι η Ευρώπη μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό. Ε, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία έτσι, δυναμικού που θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος. Το 2011 ε, δημιουργήσαμε μια κοινή στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ε, πειρατείας στη Δανία και έχουμε ένα γενικό πλαίσιο για να δούμε ποιο είναι τα θέματα ενδιαφέροντος. Βραχυπρόθεσμα, θέλουμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, ας πούμε. Ε, παραδείγματο χάρη πτήση ελέγχου και αναγνώριση, αλλά και πιο μακροπρόθεσμα δημιουργία δυναμικού capacity building, ούτω ώστε τα παράκτια κράτη να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα και κυρίω να επικεντρωθούμε στην πρόληψη τη πειρατεία. Πιστεύω ότι η διάσκεψη του Μαρτίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Δανέζικη Προεδρία θα συνεισφέρει ε, ούτω ώστε να μπει ψηλά, να τεθεί ψηλά το πρόβλημα τη πειρατεία στην ημερήσια διάταξή μα. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίω την κυρία Μάισνερ για την γνωμοδότηση πρωτοβουλία για την ε, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική του 2010, έκθεση του 2010. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι ένα κομβικό σημείο και δεν θα πρέπει να την ξεχάσουμε και στο μέλλον. Υπάρχουν ε, νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ε, θαλάσσια αυτή πολιτική και τους επόμενους μήνες θα προσπαθήσουμε ούτω ώστε να σημειώσουμε βήματα και σε αυτή την πρωτοβουλία και σε αυτό το φάκελο. Τώρα θα ήθελα να σταθώ μια στιγμή σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι αρμοδιότητά μας, δική σας και δική μου, ε, του τουρισμού, που είναι μια οικονομική δραστηριότητα μεγάλη σημασία, έχει μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, είμαστε μοναδικό τουριστικό προορισμό εδώ στην Ευρώπη και μπορούμε να προτείνουμε θαυμάσια πράγματα, φανταστικά πράγματα στου τουρίστε. Ε, αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη είναι ο πρώτο τουριστικό προορισμό σε όλο τον κόσμο. Ε, έχει μία θέση καταπληκτική και πρέπει να την κρατήσει και στο μέλλον αυτή την πρωτιά. νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε δουλειά ούτω ώστε να βοηθήσουμε τον ευρωπαϊκό τουρισμό μπορούμε, παραδείγματο χάρη, να ανταλλάξουμε γνώσει και δεδομένα για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Για να κλείσω. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την διάθεση που δείχνετε για συνεργασία και είμαι πεπισμένο ότι θα καταφέρουμε να κλείσουμε και να φτάσουμε σε όλου του απαραίτητου ε, συμβιβασμού, ούτω ώστε να βοηθήσουμε την Ευρώπη να αναπτυχθεί περαιτέρω. Είμαι τώρα στη διάθεσή σα για ερωτήσει και τώρα, αλλά και του επόμενου έξι μήνε. Σα ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Θα ακούσουμε πρώτα τους εκπροσώπους των ομάδων, τους συντονιστές. Ο κύριος Κούνα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Υπουργό που μας έδωσε μια γενική εικόνα των προτεραιοτήτων της Προεδρίας του. Σε πολλά σημεία συμφωνούμε γιατί είναι μια... Ε, αυτές οι προτεραιότητες είναι και δουλειά της Επιτροπής μας αλλά και του Κοινοβουλίου. Βασικό θέμα και λόγω της ε, ε, κατάστασης η ασφάλεια των θαλασσιών μεταφορών. Η Δανία είναι, έχει μεγάλη παράδοση στις θαλάσσιες μεταφορές και φαντάζομαι ότι θα έχει μεγάλη εμπειρία να προσφέρει στην όλη συζήτηση. Αλλά και στον ε, τομέα των, ε, ε των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης οικονομίας μπορεί να παίξει ο τομέας αυτός μια, ένα μεγάλο ρόλο. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίση χρέους, οπότε δεν θα γλιτώσει ούτε η ε, Δανία. Αν είχατε συνδέσει την ε, κορώνα σας με το ευρώ, θα έπρεπε και θα είχατε και εσείς ε, συνέπειες. Βεβαίως οι συνέπειες είναι πολλαπλές και αφορούν όλους ό,τι αφορά και, την, ε, και τα έσοδα, ειδικά όταν έχει κανείς να ε, καταβάλει σημαντικά ποσά και αυτό έχει να κάνει και με την ενεργειακή πολιτική. Νομίζω ότι από κοινού θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις ε, πλατφόρμες ε, offshore. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς ε, κατευθυντήριες γραμμές. Η θαλάσσια πολιτική είναι σημαντική και για την σωστή διαχείριση των θαλασσών μας. Αν δούμε, ας πούμε, τη Βόρεια Θάλασσα ή τη Μεσόγειο, υπάρχουν προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και χαιρετίζω το γεγονός ότι είπατε κι εσείς ότι το θέμα της ασφάλειας των πλοίων δεν είναι μόνο ε, επίκαιρο λόγο του Κώστα Κονκόρντια, αλλά ότι πρέπει να γίνει η ασφάλεια και πιο πράσινη και πιο αποτελεσματική. Βεβαίως δεν πρέπει να παραμελήσουμε ε, τι γίνεται και με τις ε, διάφορες ε, ε, ελεγχόμενες ζώνες οι οποίες έχουν να κάνουν και με διαφορετικά κριτήρια ανταγωνιστικότητας. Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την αλλαγή της σχετικής οδηγίας και πρέπει να προσέξουμε. Και πρέπει να προσέξετε και εσείς στην Κομισιό να μην υπάρξει παραβίαση των αρχών του ανταγωνισμού, στρέβλωση του ανταγωνισμού. Επίσης η ΕΜΣΑ θα παίξει σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή τη συζήτηση. Το έχει αναλάβει ο κύριος Φλέκενστάιν το θέμα αυτό ο συζητητής. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται και με την εποπτεία που θα μπορεί να έχει η ΕΜΣΑ σε τέτοιες πλατφόρμες ε, πετρελαίου ή πλατφόρμες offshore. Θα πρέπει και αυτό να το μελετήσουμε προσεκτικά. Και βεβαίω θα πρέπει να δούμε την ασφάλεια των ναυτικών εντό τη Ευρώπη. Θα πρέπει αυτό να γίνει με πολύ υψηλά πρότυπα. Το συζητήσαμε και σήμερα το πρωί για το Κώστα Κονκόρδια. Και επίση πρέπει να δούμε πώ θα μπορέσουμε όλη αυτή τη δουλειά να την κάνουμε πιο αποτελεσματικά με του περιορισμένου αυτού πόρου που έχουμε. Επίση, ε, μια ενιαία πούμε, αρχή περιπολιών. Ε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά να υπάρχει μια γενική εποπτεία. Βλέπω ο πρόεδρο ετοιμάζεται να χτυπήσει το σφυράκι του. Κλείνω, πρόεδρε. Ε, και ένα ερώτημα. Ε, Εσεί ε, την ασφάλεια μέσω του Γαλιλαίου πώ μπορείτε να την προωθήσετε, ε, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ στενά, ε, πολλά, όπως πολλά στενά σημεία περάσματα, όπως τα στενά του Γιβραλτάρ, όπως άλλα σημεία τα οποία πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά, γιατί ακριβώς εκεί είναι που διακυβεύεται πολλές φορές η ασφάλεια των ναυτικών μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλχαντράουι από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Υπουργό για την ε, εισαγωγική του ομιλία. Του εύχομαι καλή τύχη στο δανεικό εξάμεινο. Θα ξεκινήσω από το ναυάγιο του Κώστα Κονκόρδια. Κύριε Υπουργέ, είμαι και εγώ της γνώμης ότι θα πρέπει με νυφαλιότητα να διερευνήσουμε τις αιτίες αυτού του δυστυχήματος και αν χρειαστεί να θεσπίσουμε νέα μέτρα για κατάρτιση των ναυτικών, για ε, μεθόδους εκένωσης και ούτω καθεξής. Προσβλέπουμε σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά τους επόμενους μήνες. Σίγουρα η ναυσιπλοεία και οι θαλάσσιες μεταφορές συνιστούν για μας μίζωνα πρόκληση. Θέλουμε να προσελκύσουμε στο μέλλον όλο και περισσότερους νέους στον κλάδο αυτό. Γιατί υπάρχει έλλειψη εργαζομένων Άρα χρειαζόμαστε και καλή κατάρτιση και εκπαίδευση, αλλά και ελπιδοφόρες προοπτικές για τους νέους. Θα μπορούσαμε να λάβουμε πολύ άριθμες πρωτοβουλίες. Κατάρτιση εκπαίδευση των ναυτικών είναι ένα, μία μόνο πτυχή. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να υιοθετήσουμε πολύ πιο ευρεία προοπτική. Αναφερθήκατε και στην έκθεση του συναδέλφου του κ. Φλέκεστάιν για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν επικοδομητική συζήτηση και σημειώνεται κάποια πρόοδος, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια προσκόμματα στις συζητήσεις και κάποιες ε, διαφορές στις απόψεις. Για παράδειγμα, ο έλεγχος των ε, πετρελαϊκών πλατφορμών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Ναυσιπλοείας. Ποια είναι η δικιά σας γνώμη κατά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλό θα ήταν να αξιοποιήσουμε τη τεχνογνωσία, το know-how της ΕΜΣΑ, του ΕΜΣΑ και να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητές του εφοδιάζοντας τον με τις απαραίτητες εξουσίες ώστε σε περίπτωση επίγουσης ανάγκης να μπορεί να λάβει κάποια μέτρα στις ε, πλατφόρμες εξορίσεως πετρελαίου. Η, πειρατεία, σημαντική μάστιγα, οξύτατο πρόβλημα. Αναφερθήκατε σε μια διάσκεψη που θα οργανωθεί για το ζήτημα αυτό. Έχουμε και εμείς ε, συντάξει ψήφισμα για την πειρατεία και περιμένουμε με ανυπομονησία τη διάσκεψη αυτή για να λάβουμε και εμείς μέρος. Σίγουρα θέλουμε ενεργό ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Τελευταίο σημείο, τουρισμός. Φυσικά είναι πολύ ζωτικός κλάδος, αλλά από ό,τι φαίνεται λίγες πρωτοβουλίες έχουν αναλυθεί για την προώθηση του τουρισμού. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να προβλέψουμε στον κοινοτικό προϋπολογισμό μια δημοσιονομική γραμμή για να έχουμε και μια ε, χρηματοπιστωτική πολιτική υπέρ του τουρισμού. Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μας. Η κυρία Μάισνερ για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον Υπουργό για την παρουσίασή του τα... και για τα σημεία που ήθελα να θίξει για την ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα. Ήθελα εγώ να πω κάτι, όχι γιατί είμαι μόνο η ε, αλλά γιατί είναι πολύ σημαντικό και ο κύριος Κουμουτσάκος επίσης έχει αναλάβει την σχετική έκθεση. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό ένας σημαντικός τομέας αυτός, έχει δικό του τίτλο στον υπολογισμό. Και σήμερα το μεσημέρι έκανα μια συζήτηση με υπουργού από την ε, ε, Βόρεια Γερμανία και ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και μου ανέφεραν και συζήτησαν και μεταξύ τους βεβαίως το πρόβλημα που συζητάτε και εσείς για την ε, έρευνα της θάλασσας όπου τις περισσότερες φορές μιλούμε μόνο για κάποια σπάνια είδη φαλενών, αλλά πρέπει να μιλούμε όταν μιλούμε για τον τομέα αυτό και για την κατασκευή πλοίων, υψηλής τεχνολογίας πλοίων και πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις, ε, ε, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον ε, κλάδο. Η Ευρώπη τα πάει καλά μέχρι στιγμή. Έχουμε αρκετά καλή εμπειρογνωμοσύνη, έχουμε τεχνολογία την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο στι στις μεταφορέ. Γι' αυτό ρωτώ κύριε Υπουργέ, επειδή ακριβώ έχετε εσεί αυτό το κομμάτι του Υπουργείου, οι μεταφορέ και οι επιχειρήσει και η ανάπτυξη μπορούν να ε, συνδυαστούν με κάποιο τρόπο, μπορείτε να κάνετε μια επίθεση προς αυτές τις ε, πτυχέ, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε ακριβώ αυτή την ε, εμπειρογνωμοσύνη εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργήσουμε και άλλε θέσει εργασία. Και άλλο ένα ερώτημα. Ασφάλεια στι θαλάσσιε μεταφορέ. το, το αναφέρατε και εσεί. Όλοι μιλούμε για το δυστύχημα στην Ιταλία. Ε, το πρωί συζητήσαμε και με τον Επίτροπο Κάλλα. και το είπαν και οι συνάδελφοι, βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε, πρέπει να ερευνήσουμε πώς καταλήξαμε σε αυτό το σημείο. Υπήρξε ανθρώπινο λάθος, υπήρξε κάποια πράγματα που δεν ε, έτυχαν τη σωστή ε, αντιμετώπιση. Πώς μπορούμε στο μέλλον λοιπόν να δραστηριοποιηθούμε καλύτερα και και κατά τη διάρκεια της δικής σας προεδρίας. Ή έχουμε ρυθμίσει αρκετά τα πράγματα και απλώς πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τέτοια είδους, τέτοιου είδους δυστυχήματα πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε, πώς μπορούμε να καταστήσουμε τις θάλασσες πιο ασφαλείς. Επίσης, Υπάρχει μεγάλο δυναμικό ε, know-how, μεγάλη ε, εμπειρογνωμοσύνη για το πώς μπορούμε να καταστήσουμε πιο πράσινη την, ε, τις μεταφορές στη θάλασσα. Και αυτό πρέπει να το φροντίσουμε. Οπότε, ίσως να πρέπει να, να, να συνδυαστούν και κάποιες επιτροπές του Κοινοβουλίου μεταξύ τους για να δουν ακριβώς το θέμα αυτό και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Και ένα τελευταίο σημείο, το θέμα της... το θέμα της οδηγίας. μιλάμε για, ένα, ε, για μια ισότητα για, για όλες τις, ε, για αυτές τις δραστηριότητες. Ε, προφανώς πρέπει να υπάρχουν πολύ χαμηλότερες ε, αξίες θείου και πρέπει αυτό να το πετύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εσείς υπάρχει περίπτωση να προωθήσετε το θέμα αυτό γιατί είναι σημαντικό σημείο και για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος η οποία είναι επίσης σημαντική πτυχή. Ευχαριστώ κύριο Κράμερ για τους πρασίνους. Ε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε στην αρχή για τα θύματα και τις οικογένειές τους από το δυστύχημα στην Ιταλία. Δυστυχώς πέθαναν αρκετοί άνθρωποι και αυτό είναι τραγικό. Αλλά το τραγικό είναι ότι επλήγησαν και οι ακτές από τεράστιες ποσότητες πετρελαίου. Ξέρουμε ότι οι α, θαλάσσιες αυτές μεταφορές στην αυσυπλοεία χρησιμοποιούν ε, ε, μηχανές ε, καύσης χωρίς φίλτρα αέρος και συνήθως Πρέπει να, χρησιμοποιηθούν, πρέπει να γίνουν ειδικέ δηλώσει για τα καύσιμα που χρησιμοποιούν τα πλοία αυτά. Υπάρχει τώρα μία ρύθμιση για την Βαλτική, για, την, για, το θείο που, για την περιεκτικότητα σε θείο στο, στην δίζελ που πρέπει να είναι έως 0,1%. Ε, υπήρξαν κάποιες αντιστάσεις, να, υπάρξουν, ε, να υπάρξει αλλαγή των αριθμητικών στοιχείων. Θέλουμε να μας πείτε εσείς ποια είναι η θέση σας. Και επίσης, το δυστύχημα του Κονκόρντια μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως ε, κίνητρο ώστε να, επιφε... να βάλουμε κάποια όρια και για την ε, ε Μεσόγειο και για άλλες θάλασσες έτσι ώστε το, ε, τα καύσιμα που μπορεί να, μετά από ένα δυστύχημα να βγουν στη θάλασσα να μην είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Μπορεί να, αυτό να σημαίνει αύξηση του κόστους, αλλά σημαίνει όμως ότι θα υπάρξει μεγαλύτερο όφελος για την ναυσιπλοεία. Δεύτερον, και σε σχέση μάλλον με αυτό, ε, ακριβώς επειδή αυτά είναι, τα πλοία είναι κρουαζιερόπλια, η Ένωση Προστασίας της Φύσης ε, θεώρησε ότι ε, η, τα κρουαζιερόπλια ανήκουν στην αεροπλοεία και όχι στην αυσιπλοεία γιατί κάνουν πολύ μεγάλα, έχουν πολύ μεγάλα κέρδη και εκπέμπουν πάρα, πολύ, πάρα, πολλές, πάρα πολλά καυσαέρια. Ερώτημα λοιπόν, εσείς στην Προεδρία σας θα φροντίσετε ώστε να υπάρξει, να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει για το, για το δυστύχημα της Ιταλίας, αλλά να δούμε τι θα γίνει και με τα δεξαμενόπλια διπλού κήτους και γενικά με όλα τα σκάφη που χρησιμοποιούν τέτοια βαριά καύσιμα. Υπάρχουν ε, στην ε, Ευρώπη πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά σημεία, κυρίως στην ε, Βαλτική, τα οποία είναι όντως κομμάτια σημαντικά από τα οποία περνούν πλοία και τα οποία θα πρέπει να ενταχθούν στο, στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, μπορεί να είναι το κόστος ε, αρκετό, αλλά ε, είναι πολύ σημαντικό να μπουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ξέρετε ότι οι τουρίστες περνούν από πολλά σημεία και ο τουρίστας με το που κάνει μια κρουαζιέρα θα δώσει πολύ περισσότερα χρήματα στην τοπική κοινωνία από έναν τουρίστα που περνάει απλώς με το αυτοκίνητό του και διέρχεται από κάποιες περιοχές. Επίσης, η στρατηγική της Βαλτικής που είναι ανεξάρτητοι από τα διάφορα, μέλη, ε, τα διάφορα κράτη, είτε είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε όχι. Αυτή η στρατηγική σημαίνει ότι όταν κάποια κράτη συνεργάζονται μπορούν να υποφεληθούν. Υπάρχει στρατηγική για το Δούναβι. Δέκα κράτη ε, τα αφορά αυτή η στρατηγική. Για τη Μεσόγειο επίσης μπορούμε να δούμε ότι όταν τελικά ε, συνδυάζουμε τις δυνάμεις μας ε, μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα από ό,τι όταν βρίσκεται ο ένας απέναντι στον άλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και περιμένω την απάντηση. Η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη από τον Υπουργό που δεν πρόλαβα να έρθω νωρίτερα. Αλλά ευτυχώ ήταν εδώ ο βοηθός μου και κράτησε σημειώσεις από την ομιλία σας συμφωνώ με τους συναδέλφους για τα πρωινά επί... σχόλια του Επιτρέπου σε ό,τι αφορά τραγικό δυστύχημα του Κονκόρδια στις Ιταλικές ακτές. Ε, το συζητήσαμε εκτενώς και με τον Επίτροπο το πρωί. Φυσικά εσείς ως Δανική Προεδρία θα διαμορφώσετε και τη δική σας γνώμη. Περιμένουμε λοιπόν ε, την έκβαση της έρευνας και αν χρειαστεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα είτε από τον κλάδο είτε από το κοινοβούλιο ή από άλλο θεσμικό όργανο. Περιμένουμε συνέχεια. Κρατήσαμε πάντως σημειώσεις από αυτά που μας είπατε και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με τη Δανική Προεδρία κατά το εξάμεινο αυτό. Βέβαια, στη δική σου εντολή περιλαμβάνεται και η οικονομική μεγέθηση και οι επιχειρήσεις, γιατί όλοι χρειαζόμαστε και οικονομική ανάπτυξη και ε, άθηση των επιχειρήσεων και οι μεταφορές θα παίξουν ζωτικό ρόλο σε κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε ρυθμίση, αλλά όχι παντού, όπου όντως προσφέρει κάτι. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως θα πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική ρύθμιση. Ε, στον τουρισμό, στις μεταφορές είναι σημαντικό η Ευρώπη ως Ήπειρος να έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης. Και αυτή η ανάπτυξη να ωφελήσει όλα τα κράτη-μέλη και όχι ορισμένους επίλεκτους μόνο. Ευχαριστώ κύριε Σκόχλιτσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, ελπίζω ότι η Ιδανική Προεδρία θα καταφέρει να διερευνήσει ε, διεξοδικά το, το δυστύχημα στις ιταλικές ακτές του Κώστα Κονκόρδια και περιμένουμε τα πορίσματα αυτής της έρευνας. Δεύτερον, τι πρόοδος υπάρχει σε ό,τι αφορά τα παλιά δεξαμενόπλια. Γιατί τα παλιά δεξαμενόπλια της Ευρώπης εξάγονται και παροπλίζονται ή διαλύονται στην Αφρική ή σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτο ερώτημα, πλωτές μεταφορές, ποτάμιες μεταφορές. Σημαντικός τομέας, γιατί και οι πλωτές μεταφορές είναι σημαντικές ως ξεχωριστή κατηγορία για την ανάπτυξη του τουρισμού. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θέλετε να απαντήσετε πρώτα στους συντονιστές και μετά να περάσουμε στον τρίτο γύρο με τους πέντε ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ για τα σχόλια και για, και τις πολύ επικοδομητικές σας ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά που υπόθηκαν οι ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε την κατάρτιση των ναυτικών, εκπαίδευση των ναυτικών. Στο Συμβούλιο εξετάζουμε κάποιες τροπολογίες. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι χρειάζονται νέα μέτρα. Πάντως η Προεδρία θα επιδιώξει συμβαστική λύση και συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα όμως μας ενδιαφέρει ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να υπάρξει κατανόηση των διαφόρων θέσεων. Η Ιδανική Προεδρία θα αφιερώσει όσο χρόνο χρειάζεται στην ε, ανέβρεση συμφωνίας που θα καλύπτει και το θέμα της κατάρτισης των ναυτικών. Το θέμα της οδηγίας για το θείο και ε, αυτό το ζήτημα αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, επικαιροποιήσει τη συμφωνία, την οδηγία για το θείο, ώστε η, η διατάξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυσιπλοείας ε, να περιληφθούν και στο κοινοτικό δίκτυο. Και υπάρχει και το θέμα της γαλάζιας ανάπτυξης. Μπορεί να είναι χρήσιμο αυτό το εργαλείο για την η φόρο ανάπτυξη της ναυσιπλοείας και των θαλάσσιων μεταφορών. Αλλά η μπλε ανάπτυξη είναι μόνο μία εναρκτήρια φάση, μία φετηρία. Στο μέτρο που θα αναπτυχθεί περαιτέρω αυτή η πρωτοβουλία, θα εξασφαλίσουμε μια πραγματικά φόρο ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών και ίσως ε, αυξηθούν και οι κοινοτικέ αρμοδιότητες στον τομέα αυτό. Μα ρωτήσατε ποια είναι η θέση της Δανικής Προεδρίας σε ό,τι αφορά τον ε, σχεδιασμό των θαλάσσιων μεταφορών, τον προγραμματισμό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εθνικές αρμοδιότητες για τη χωροταξία κατά κάποιο τρόπο στις θάλασσες. Έχουμε πάντως μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία τη ευρωπαϊκή Επιτροπή που οριοθετεί κάπως ε, τα πράγματα, το πλαίσιο για το τι ρύθμιση επιτρέπεται στη χωροταξία αυτή, στη θάλασσα, ε, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και το περιβάλλον, η προστασία του περιβάλλοντος. Δεν ξέρω πάντως αν θα προλάβουμε στη διάρκεια της ε, Δανικής Προεδρίας να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Σχεδόν όλοι οι ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στο δυστύχημα του Κώστα Κονκόρντια. Αυτό το ναυάγιο, αυτό το δυστύχημα μας βάζει σε σκέψεις και προβληματισμό, κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και περιμένουμε την έρευνα για τη βήθηση του πλοίου και όπως είπε και ο Επίτροπος Κάλλας, με βάση τα απορίσματα της έρευνας θα δούμε τι ε, μέτρα και τι διατάξεις χρειάζονται για να ενισχύσουμε την ασφάλεια και των επιβατικών πλοίων και των επιβατών και των ναυτικών. Πρώτα απ' όλα όμως περιμένουμε τη διεξοδική έκθεση για τις συνθήκες του δυστυχήματος και για τις συνέπειες του. Μόνο μετά θα κληθούμε να λάβουμε απόφαση για θέσπιση ενδεχομένω νέων κανόνων βλέποντας και κάνοντας ως προς το Κώστα Κονκόρδια και τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Σε ό,τι αφορά την οδηγία STCW, Διεθνή Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευση Έκδοση Πτυχίων και Τήρηση Φυλακών των Ναυτικών. Το δυστύχημα του Κώστα Κονκόρδια μας έδειξε πόσο άμεση επιτακτική ανάγκη υπάρχει για την συμπερίληψη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των διατάξεων αυτής της Διεθνούς σύμβαση για τα Πρότυπα εκπαίδευση. Ε, ναυτικών. Θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την ε, ενσωμάτωση στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο της Διεθνούς Αυτής Σύμβασης, STCW. Επίσης, ε, πολλοί μίλησαν για τις αρμοδιότητες ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας και των σχετικών συμβάσεων για την εργασία των ναυτικών. Θα πρέπει να εγκρίνουμε, να κυρώσουμε αυτή τη διεθνή σύμβαση για τις εργασίες στη θάλασσα για να τεθεί σε το ταχύτερο σε εφαρμογή και να εξασφαλίσουμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες και καλύτερη, μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ναυτικούς. Φυσικά λαμβάνοντας υπόψη και το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Σε ό,τι αφορά τα δεξαμενόπλια τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ρυθμίση και για τις offshore πλατφόρμες Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ασφάλεια των πλατφορμών αυτών ε, offshore. Ήδη υπάρχουν αυστηροί κανόνες σε πολλά κρατημέλη που διαθέτουν τέτοιες ε, ε, υπεράκτιες πλατφόρμες εξόριξης πετρελαίου. Μία άλλη ερώτηση αφορούσε την πειρατεία. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση της πειρατείας είναι προτεραιότητα πολλών χωρών και θεωρώ ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναμειχθεί ενεργά στη συζήτηση αυτή και να συμμετέχει στην ανέβρεση λύσεων για την αντιμετώπιση της, θερα... της πειρατείας που αποτελεί μάστιγα της ναυσιπλοείας. Αναφέρθηκε και ο τουρισμός. Στον τριμερή διάλογο, ε, μάλλον στο τρίο των προεδριών, οι τρεις διαδοχικές προεδρίες Πολωνίας, Δανίας και Κύπρου ε, εξέτασαν αυτό το θέμα, αλλά δεν ε, έχουμε προγραμματίσει ειδικέ διασκέψεις για τον τουρισμό στη διάρκεια της ιδανική Προεδρία. Είναι σαφές πάντως ότι και ο τουρισμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κοινοτικών πολιτικών και θα προωθεί με διάφορες πρωτοβουλίες ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τονωθεί η εσωτερική αγορά και να εξασφαλίσουμε παρόμοιες συνθήκες παντού και ε, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ε, του ευρωπαϊκού τουρισμού. Η κυρία Μάισνερ μίλησε για την έρευνα. Και είπε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα η έρευνα, η ε, πόρη και η τεχνογνωσία που διαθέτουμε στις θαλάσσιες μεταφορές. και στα πλαίσια του Κώστα Κονκόρδια επαναλαμβάνω ότι ας περιμένουμε πρώτα την έρευνα και τη διαλεύκαση του δυστυχήματος ε, και μετά να δούμε αν θα πρέπει να θεσπίσουμε επιπλέον μέτρα. Η κυρία Μάισνερ έθεσε και την ερώτηση των πράσινων θαλάσσιων μεταφορών. Πραγματικά αυτό το θέμα είναι συναρπαστικό ιδιαίτερα για μας τους Δανούς που αναζητούμε και εναλλακτικά καύσιμα που θα αντικαταστήσουν τα κλασικά καύσιμα. Γιατί όχι φυσικό αέριο, γιατί να μην κατασκευάσουμε κινητήρες που να λειτουργούν με φυσικό αέριο. Στη Δανία γίνονται έρευνες για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για το θείο, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, εμπίπτει περισσότερο στις αρμοδιότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος. Πάντως, ο Υπουργός Περιβάλλοντος ε, ευελπιστεί ότι θα διεκπαιρεώσει τις διαπραγματεύσεις ε, της οδηγίας αυτής στη διάρκεια του δανεικού εξαμήνου. Ο κύριος Κράμερ ε, ρώτησε τι θα γίνει με τη στρατηγική για τη Βαλτική. Δεν υπάρχει σαφή στρατηγική για τη Μεσόγειο, αλλά αν υποβάλει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα την εξετάσουμε πολύ ευχαρίστως. Κυρία Φώστερ, ε, ευχαριστώ θερμά για τις ε, παρατηρήσεις σας και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο θέμα του αθέμητου ανταγωνισμού που μερικές φορές διαπιστώνουμε στην Ευρώπη. Και πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη είναι το ζητούμενο και σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε όμως πρώτα να βρούμε μια λύση ε, για το χρέος, το υπερβολικό χρέος ορισμένων χωρών και να διορθώσουμε την κρίση στην Ευρωζώνη δίνοντας νέα όθηση στην ανάκαμψη. Νομίζω ότι δίνοντας έβαση στην ανάκαμψη θα εξέλθουμε πιο εύκολα από την κρίση και του χρέους. Σε ό,τι αφορά τώρα την ολοκλήρωση των διαφόρων διαδρόμων, ευρωπαϊκών διαδρόμων. Αν κατάλαβα καλά, ε, είπατε ότι τα προγράμματα αυτά δεν θα πρέπει να τύχουν ειδικού προϋπολογισμού, αλλά να υπάρχει ένα γενικό κονδύλιο. Στη Δανία δεν έχουμε πολλούς ε, ε, περιφερειακούς δρόμους, αλλά φαντάζομαι άλλες χώρες έχουν πολύ περισσότερους και τους ενδιαφέρονται για μια συζήτηση για τους περιφερειακούς αυτούς δρόμους. Αυτά και ελπίζω να απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Τέσσερις ακόμα μιλητές έχουν ζητήσει το λόγο, οπότε θα τους δώσουμε το λόγο και μετά θα απαντήσει και πάλι ο Υπουργός. Ο κύριος Ρίκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την ε, παρουσία σας. Καλή τύχη για τους επόμενους 6 μήνες. Ε, η Δανία με μεγάλη χαρά έχει έναν Υπουργό Ανάπτυξης. Ε, τη, σήμερα ημέρα είναι πολύ σημαντικό ένας Υπουργός Ανάπτυξης. Τέσσερις ερωτήσεις. Ε, οι τρεις πρώτες, ε, επειδή είστε υπεύθυνο για την ανάπτυξη και για τις επιχειρήσεις. Πάνω στο γραφείο της ε, Προεδρίας υπάρχει ένας φάκελος σημαντικός για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τη χρηματοδότησή τους. Φυσικά, διάφοροι συνάδελφοι στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, Περιφερειακή Επιτροπή, έχουν ε, τις απόψεις. Εγώ θέλω να πείτε την άποψή σας. Ε, επειδή είστε υπεύθυνο για την ανάπτυξη, έχω να σας πω ότι ακόμα και οι οίκοι βαθμολόγησης ε, ανησυχούν για την ανάπτυξή μας, οι οίκοι βαθμολόγησης πιστολιτικής μας ικανότητας εννοώ, ανησυχούν για την ανάπτυξή μας, γιατί θεωρούν ότι το παρακάνουμε τη λιτότητα. Τι πιστεύετε για το ποσό που προτείνετε, που είναι 50 δισεκατομμύρια, ε, συνολικό ποσό είναι αυτό, είναι σωστό ποσό ε, στα πλαίσια της επόμενης περίοδου του επόμενου, της επόμενης πολιετής ε, περίοδου περίοδου. Προτιμάτε τις επιδοτήσεις επίσης ή όχι. Και επίσης για τα ομόλογα έργων. Ποια είναι η προσωπική σας άποψη. Ε, Επίση, μια τέταρτη ερώτηση για τα θαλάσσια θέματα. Κάθε φορά που υπάρχει ένα θαλάσσιο ατύχημα, όποιο και αν η φύση του, πάντα ε, ε, σκεφτόμαστε πώς θα αδειάσουμε τις δεξαμενές των, από τα καύσιμα. Ε, εδώ υπάρχουν 250... 2,5 νομίζω χιλιάδες τόνους καύσιμα. Κάπως θα πρέπει να τα αδειάσουμε. Υπάρχουν μηχανισμοί για να μπορέσουμε να διάσουμε τα πετρελαϊκά προϊόντα γιατί η δυνατότητα να φτάσουμε στις δεξαμενές ε, των πλοίων όταν υπάρχει ε, καταστροφή είναι δύσκολη. Είναι μικρές αυτές οι δυνατότητες. Το υπάρχει ένας μηχανισμός ε, που δεν είναι πολύ ακριβώς και που μας επιτρέπει σε περίπτωση ατυχήματος να φτάσουμε στις δεξα... δεξαμενές των πλοίων και να διάσουμε, να διάσουμε τα καύσιμα. Ε, πιστεύετε ότι έχει νόημα να έχουμε αυτόν το μηχανισμό. Προς το παρόν δεν γίνεται τίποτα. Ενώ υπάρχει αυτή η λύση. Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός. Αυτός ο εξοπλισμός. Ο κ. Ουτζίας. Πώς θα πούμε τον Πονηφικά. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ Οικονομικής Ανάπτυξης. Όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Ρικέ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Επιτρέψτε να είμαι ειλικρινή μαζί σα. Θέλω να σας μιλήσω για την απογοήτευσή μας για το πρόγραμμα που αφορά τον τουρισμό. Μήπως ε, σας διέφυγε κάποια από τις σελίδε που είχατε τις ομιλία σας και δεν την... Ε, γι' αυτό δεν αναφέρατε τίποτα. Ποιε είναι οι προθέσει τη Δανέζικη Προεδρία για τον τουρισμό, γιατί μα είπατε κουβέντα. Ε, περιμένουμε πολλά από την πολιτιστική μας και τουριστική μας κληρονομιά στην Ευρώπη. Δηλαδή μπορούμε να πετύχουμε και ανάπτυξη και χάρη στον τουρισμό. Σας παρακαλώ θερμά να λάβετε υπόψη σας αυτή την έκκληση που σας εκφράζω. Δύο σκέψεις θέλω να εκφράσω για το ζήτημα του, της τραγωδίας του Κώστα Κονκόρντια να σας υπενθυμίσω ότι το, η τραγωδία αυτή του Κώστα Κονκόρντια δεν είναι η μοναδική πρόσφατη τραγωδία που έπληξε τον τομέα των κρουαζιερόπλοιων. Μην ξεχνάτε ότι πριν από δύο χρόνια, όχι στη Μεσόγειο όμως, ένα ολόκληρο πλοίο ε, επλήγει από μία καταιγίδα και είχε 800 επιβάτες, το αποτέλεσμα είναι, ήταν πάρα πολλά θύματα. Για να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα, τέτοια ατυχήματα, ε, για να μην ξαναγίνει κανένα ατύχημα, ίσονο, πιο ίσονο ε, σημασίας. Στις ακτές της Ισπανίας, θα θυμάστε, πέρυσι, ε, τι συνέβη ένα άλλο ατύχημα με ένα άλλο Κουρασγερόπουλιο. Και άλλου τύπου τέτοια ατυχήματα έχουν ξανασυμβεί. Σήμερα το πρωί, στο συναδελφό σα για τι μεταφορέ, ε, είχα τονίσει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διάσταση, με το μέγεθο αυτών των πλοίων και με τον αριθμό των επιβατών που φέρουν. Ε, είναι ολόκληρα παλάτια, είναι ολόκληρα ολόκληρε πολυκατοικίε με δεν ξέρω και εγώ πόσου ορόφου και είναι δύσκολο να τα διαχειριστούμε αυτά τα πλοία. Ο κύριο Ρικέ έθεσε ένα ερώτημα Μην ξεχνάτε ότι το Κώστα Κονκόρδια, επειδή είχε αυτό το σχήμα, ε, με το που έγειρε, ξαφνικά όλα τα ηλεκτρικά συστήματα παρέλυσαν. Ε, γιατί? γιατί όλα τα ηλεκτρικά συστήματα, η, λειτουργία τους ας πούμε, ρυθμιζόταν ε, σε ένα πάτωμα πολύ κοντά στη θάλασσα. Μήπως θα πρέπει να τα βάλουμε πιο ψηλά όλα αυτά τα, τα μηχανήματα για να μην βρέχονται και αμέσως παραλύουν. Ε, Μήπω θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ε, ένα κανονισμό για το θέμα αυτό και ζητώ συγγνώμη που τα λέω έτσι έξω τα δόντια, ειδικά για το θέμα του τουρισμού. Ε, αλλά επειδή σας ξέρω ότι είστε ευαίσθητος άνθρωπος, ξέρετε ότι. Ε, εντάξει, μετά, μετά από λίγο θα σας περάσει αυτή η ταραχή που σας προκάλεσα. Ο κ. Κουμουτσάκος. Thank you, Chair. Um, thank you, uh, thank Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την έμφαση που δίδατε σε αυτό το θέμα της αντιμετώπισης της πειρατείας. Η πειρατεία πραγματικά έχει γίνει ένα μια επιχείρηση χαμηλού κινδύνου και υψηλού κέρδους ειδικά για την ε, σταθερότητα του παγκοσμίου εμπορίου, των ε, θαλασσιών μεταφορών. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, ζήτημα και θα πρέπει να το δούμε. Ιδιαίτερα να σκεφτείτε ότι το ετήσιο κόστος για την παγκόσμια οικονομία λόγω της πειρατείας φτάνει τα 7 με 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Από την άλλη βλέπουμε ότι από το 2009 ο ρυθμός των πλοίων στις ε, ε, αποστολές ε, ΝΑΦΟΡ έφτασε από τα 35 τα 10 και αυτά τα 10 συνήθως συνοδεύουν πλοία του Παγκοσμίου Προγράμματος Επιζητισμού του ΟΗΕ. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ποια είναι η ευρωπαϊκή παρουσία μας στην περιφέρεια. Περιμένουμε λοιπόν την διάσκεψη που θα οργανώσετε με την Κομισιόν στις 28 και 29 Μαρτίου, όπως είπε και ο συνάδελφος Αλχαντράουι, ε, και εμείς περιμένουμε να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου σε αυτή τη διάσκεψη. Και να σας πω επίσης ότι κατά πάσα πιθανότητα ως συνέχεια της πρωτοβουλίας που λάβαμε με τον, ε, αποκοινούμενο Βαντάλεν, θα κάνουμε μια συζήτηση μετά από μια προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου κατά πάσα πιθανότητα, στο Στρασβούργο. Ή μάλλον το Μάρτιο. Οπότε περιμένουμε την παρουσία της Προεδρίας σας και την ενεργό συμμετοχή της σε αυτή τη συζήτηση. Και βεβαίως ελπίζω ότι και η Κυπριακή Προεδρία θα ακολουθήσει τις ε, προσπάθειες που κάνετε σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για τα συλληπιτήριά σας ε, για το ατύχημα του Κονκόρδια, του Κώστα Κονκόρδια. Και θέλω να συμφωνήσω με αυτά που είπατε στην ε, ομιλία σας. Ε, πηγαίνω προ προς την ίδια κατεύθυνση με αυτά που είπε σήμερα το πρωί ο Επίτροπος Κάλλας. Έχετε μια προσέγγιση κι εσείς πολύ ρεαλιστική και ισορροπημένη. Κύριε Κόλετσεκ, ε, έχετε, έφυγε ο κ. Κόλετσεκ στο μεταξύ, αλλά θέλω να σας πω ότι οι έρευνες είναι ακόμα εν εξελίξη για να δούμε ποιες είναι οι ποινικέ και αστικές ευθύνες. Ε, Φυσικά θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει το ρόλο της, αλλά μην νομίζετε ότι οι Ιταλικές Αρχές κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Κάνουν ό,τι προβλέπεται από τον νόμο, ούτω ώστε ε, να μαθευτεί η αλήθεια ε, προς όφελος όλων της Ιταλίας, ε, της Ευρώπης, η τεχνική και ε, ανθρώπινη αλήθεια. Και ποινική, ε, ή μάλλον δικαστική αλήθεια. Θα είμαι πιο ειλικρινής από τον κύριο Τζίας για τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το, το πρόγραμμα COSME υπέρ της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και παρατήρησα ότι είναι ένα πρόγραμμα που η Δανέζη και η Προεδρία θεωρεί προτεραιότητας. Ε, στο εσωτερικό προβλέπεται ένα κονδύλι για να υποστηρίξουμε την πολιτική τουρισμού 131 εκατομμύρια ευρώ για 7 χρόνια με βάση την πρόταση της Κομισιόν. Λίγο-λίγο στο εσωτερικό του Συμβουλίου δημιουργείται μια ε, πολεμοχαρής ε, ε, ομάδα χωρών που θεωρούν ότι δεν πρέπει να προβλέψουμε κονδύλια για να υποστηρίξουμε αυτές τις, αυτή την πολιτική πέρα από αυτά που κάνει το Κοινοβούλιο, γιατί το Κοινοβούλιο εκφράστηκε με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ τη δέσμευση για μια οικονομική στήριξη για την πολιτική τουρισμού, σα ρωτάω από πλευρά δική σα Προεδρία, πέρα από τι διασκέψει λοιπά που προφανώ έχουν το, τη σημασία του, αλλά εσεί δεσμεύεστε ω Προεδρία ε, για να κάνετε ό,τι μπορείτε, ούτω ώστε να ξεπεράσουμε αυτή την έχθρα των, αυτών των κρατών μελών και για να προστατεύσουμε αυτόν τον μικρό θησαυρό των 131 εκατομμυρίων. Εγώ δεν λέω να τον αυξήσουμε, αλλά όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο τουρισμός είναι σημαντικό τομέα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα όλη τη Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Φιντάντζα. Ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Υπουργέ, αν μπορώ και εγώ να σας υποβάλω για το θέμα της πειρατεία. Η πειρατεία ίσως θα πρέπει να αλλάξει ακόμη και ως όρος, γιατί οι περισσότεροι ε, όταν ακούνε πειρατέ, φαντάζονται τον Τζόνι Ντεπ μέσα σε ένα μεγάλο πλοίο και στα μέσα της ε, ταινία τη γνωστή. Ε, οι πειρατέ συνήθω δεν είναι τόσο ευγενεί όπω ο Τζόνι Ντεπ, είναι εγκληματίε. Νομίζω ότι πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε λίγο και την αντίληψη που έχουμε για τους πειρατέ. Αυτό που έχει βεβαίω μεγάλη σημασία είναι η μείωση τη ε, δύναμη τη ΝΑΦΟΡ στην ΝΑΦΟΡ τη ε, Ευρώπη. Ε, πρέπει να δούμε πώς θα οργανωθούν και οι υπόλοιποι στόλοι για να συντονίσουμε και εμείς την έρευνα για την έβρεση αυτών των ανθρώπων και πρέπει να δούμε ποιε είναι οι δράσει που θα αναλάβουμε σε περίπτωση που υπάρξει προσπάθεια κατάληψης ενό πλοίου Ίσως να μπορούν να μας δώσουν τα βασικά πλοία η Ηνωμένο Βασιλείο, Γαλλία και η ΕΠΑ. Αλλά δυστυχώ έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει ένα μεταγωγό ε, πλοίο και πρέπει να υπάρχουν και κάποια πλοία γύρω-γύρω του για να το βοηθούν. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η ΝΑΦΟΡ ε, αποτελεσματική. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανησυχία εδώ στο Κοινοβούλιο ότι η ΝΑΦΟΡ δεν έχει τους πόρους που χρειάζεται για την περιοχή που πρέπει να καλύψουν. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε από την τελευταία ερώτηση. Το θέμα της πειρατείας δηλαδή. Χαίρομαι που και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και η Προεδρία μα θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα η καταπολέμηση αυτού του είδους εγκληματικότητα. Πρόκειται για μια άγρια και βίαιη εγκληματικότητα. Γιατί... Μιλάμε <coughs> για ένα τομέα που ε- εκμεταλλεύονται και κάνουν πανηγύρι οι εγκληματίες. Όπω είπατε κι εσεί είναι μεγάλη απειλή εναντίον των θαλάσσιων μεταφορών, αλλά και εναντίον των ναυτικών των ίδιων. Και εμείς ως Προεδρία θέλουμε να σα πούμε ότι δεσμευόμαστε, ούτω ώστε να γίνει μια διεθνή συντονισμένη προσπάθεια κατά τη πειρατεία και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην, στα πλαίσια της διεθνούς προσπάθειας που γίνεται και για το capacity building, και για να υπάρξει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Έχουμε αυτή τη διάσκεψη που οργανώνουμε και χάρη σε αυτή πιστεύουμε να συνεισφέρουμε κι εμείς στο να πλαισιώσουμε αυτό το θέμα και να διευκολύνουμε ένα διάλογο πιο στενό με το Κοινοβούλιο. Πολλοί από εσά μίλησαν επίσης για τον τουρισμό. Για το σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια τα οποία έχουν ακουστεί. Φυσικά, ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για την Ευρώπη και για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Και το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι ένας από τους μεγαλύτερους ε, τουριστικούς προορισμούς θα πρέπει να μας ε, κινητοποιήσει για να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτή την οικονομική δραστηριότητα. Εγώ στην παρέμβασή μου δεν είπα ότι θα υπάρξει προτεραιότητα στον τουρισμό, όντως. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να μελετήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Να δούμε ποια στοιχεία αποτελούν τμήμα της ενίας αγοράς και μπορούν να συνεισφέρουν ε, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μας εμείς και η επόμενη Προεδρία, η Κυπριακή αλλά και η προηγούμενη Πολωνική, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε στην ατζέντα τον τουρισμό. Τον Ιούνιο του 2010 έγινε μια ανακοίνωση της Επιτροπής για τον Τουρισμό με 21 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε τέσσερις τομείς. Ε, Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού, ε, βιώσιμος τουρισμός, βελτίωση της εικόνας της Ευρώπης, σαφείς ε, ευθύνες, ε, ποιοτική τουριστική προορισμή και σωστή χρήση των ε, οικονομικών μέσων. Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες αυτές που έχουν διατυπωθεί έχουν ήδη ξεκινήσει, έχουν δρομολογηθεί. Και έχουμε την εντύπωση ότι η Κομισιόν έχει αρχίσει τη μελέτη πολλών άλλων πρωτοβουλειών για τον τουρισμό και ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα εμπλακούν, θα δώσουν τη γνώμη τους σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του τουρισμού. Φυσικά θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι Απάντησα στην πρώτη και τελευταία ερώτηση. Ε, τώρα, για την πρώτη ερώτηση για τις, α, τους πόρους για τις υποδομές. Αυτό δεν είναι η άμεση αρμοδιότητά μου, είναι ε, αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών. Αλλά τα κονδύλια για τις υποδομές θα πρέπει να τα δούμε και να τα εγγράψουμε στο γενικό προϋπολογισμό. Εμείς ε, τονίζουμε ότι η ποιότητα και η αριστεία είναι βασικά στοιχεία για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πόρους για τις υποδομές. Αλλά όπως σα είπα, ο συνάδελφός μου Υπουργό Οικονομικών ασχολείται με το θέμα αυτό. Μιλήσαμε επίση για τα project bond, για τα ομόλογα έργων. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το θέμα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά και αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών. Πολλέ ερωτήσεις και παρατηρήσει. Ακούστηκαν για την θαλάσσια καταστροφή, για το Κώστα Κονκόρδια. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ασφάλεια, σε όλες τις πτυχές ασφάλειας. Και αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα μόνο όταν ε, μάθουμε τις, αιτίες, τις αιτίες του ατυχήματος αυτού. Μόνο τότε θα καταλάβουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τους κανόνες, τους βελτιώσουμε για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια Μπορούμε να δούμε τι γίνεται και με τα πλοία ε, διπλοκή του. Εξάλλου είναι στο τραπέζι για τη διαπραγμάτευση και ελπίζω να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό το σημείο αυτό. Ακούσαμε κάποιες ερωτήσεις. Για τα καύσιμα αλλά νομίζω ότι σας, απαντήσαμε στα καύσιμα στις προηγούμενες, ε, στο προηγούμενο γύρο απαντήσεων. Τα καύσιμα για τα ακροασγερόπλια είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό που να δούμε αν μπορούμε να έχουμε καλύτερα, λιγότερο μολυσματικά καύσιμα. Λιγότερο υπογόνα. Και επίσης είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να διάζουμε τις ε, δεξαμενές για να αποφύγουμε μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές όπως αυτές στο παρελθόν. προγραμματιάσμα λοιπόν τη δεξαμενή των καυσίμων. Πολύ σημαντικό. Τώρα, οι τελευταίε ερωτήσει που ακούστηκαν. Η μία ήταν για τη διάσκεψη. Α, μου είπατε ότι πρέπει να συμμετάσχω στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Χαίρομαι για αυτή την πρόσκληση και σίγουρα θα είναι σημαντική η παρουσία μου ε, με βάση τις ε, αρμοδιότητες που έχω. Το πρόγραμμα COSME. Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας θα ασχοληθεί με αυτό και θα το συζητήσει αυτό το σημείο. Θα το θα επιληφθεί στο Συμβούλιο Μαΐου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Υπουργέ, για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ που απαντήσατε σε ερωτήσεις των βουλευτών. Περιμένουμε την εποφελή συνεργασία μαζί σας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Όπως είπα και στους αδέλφους νωρίτερα, θέλουμε να συνεργαστούμε εκ του με την Προεδρία για να προχωρήσουμε τους φακέλους, για να σας βοηθήσουμε στη δουλειά σας, στην προσπάθειά σας είμαστε εδώ. Για να σας διευκολύνουμε. Και ελπίζω ότι θα σας ξαναδούμε μετά τη Δανέζικη Προεδρία, όταν κλείσει για να μας κάνει ένα απολογισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και περιμένουμε να σας ξαναδούμε και στο μέλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω κλείνοντας που, μου αποθύνετε αυτή την πρόσκληση, που με δεχτήκατε εδώ στην Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας, πολύ επικοδομητικές. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Αυτές οι συναντήσεις είναι πολύ σημαντικές για την Προεδρία, γιατί μας επιτρέπουν να εξασφαλίσουμε στενό διάλογο για να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, όλα τα θέματα που υπάρχουν στην ατζέντα μας. Σας υπόσχομαι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ολοκληρώσουμε όσο περισσότερους φακέλους γίνεται και σας ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις σας. Θα τις λάβω όλες υπόψη.